Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Letzter Sitzungstag der Sommerpause. Καλημέρα. Καθίστε για να ξεκινήσουμε την τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Κρίμα που δεν τα κατάφεραν όλοι να είναι παρόντες για την αρχή της συνεδρίασης. Έχουμε μια παρουσίαση μια έκθεση ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου Η πρώτη με την οποία ξεκινάμε είναι η έκθεση παρελθόν 8 του 2017 για τον έλεγχο της αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Γιάννος Βοχεζόφσκι. Και σας δίνω το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τη χαρά να παρουσιάσω uh, Uh, e ε, έχω τη χαρά να ε, παρουσιάσω στην Επιτροπή το σχέδιο γνωμοδότησης για τον έλεγχο της ε, αλίας. Όπως γνωρίζετε, η στόχος της πολιτικής αυτής είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος και αυτό ακριβώς υπήρξε και το αντικείμενο του ελέγχου μας και το ερώτημα, το ελεγκτικό ερώτημα που ετέθη. Θέλω να σας δείξω την παρουσίασή μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Λοιπόν, θα συνεχίσω, γιατί κάποια τεχνικά προβλήματα υπάρχουν. Το ερώτημα του ελέγχου ήταν, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της αλίας. Και το τα θέματα που ε, εξετάσαμε ήταν στοιχεία για το στόλο, ήταν τα, οι κυρώσεις, οι επιθεωρήσεις ελέγχθηκαν ε, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με έμφαση στη Σκοτία. Και η απάντηση στην ερώτηση μετά τον έλεγχο είναι, στην ερώτηση αν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απάντηση είναι όχι ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα επαρκώς αποτελεσματικό σύστημα για τον έλεγχο της αλίας. Έχει σημειωθεί πρόοδος τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρά τα αυτά τα κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως τον ε, κανονισμό του ελέγχου. Κάποιες διατάξεις του κανονισμού πρέπει να τροποποιηθούν. Τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής. Πρώτον, είναι θέμα στοιχείων του ε, στόλου, τα οποία δεν είναι αξιόπιστα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του καταγεγραμμένου στόλου των κρατών μελών ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή υπάρχουν σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στα κράτη-μέλη και όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντιστρόφως. Αυτό ε, και εν γέννη αυτό το μητρό του στόλου δεν είναι πλήρες και αξιόπιστο. Συνιστούμε να ε, ε, θεσπιστούν διαδικασίες για την επαλήθευση της πληροφορίας όσον αφορά το, το Μητρό Στόλου, αυτό αφορά τα κράτη-μέλη και όσον αφορά την Επιτροπή, η επαλήθευση του, ε, της δυναμικότητας και της ισχύω του κινητήρα. Τώρα, το δεύτερο συμπέρασμα αφορά τα μέτρα διαχείρισης, κυρίως τα συστήματα παρακολούθησης των σκαφών. 89% του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι συνδεδεμένο την με το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού. Ε, ένα μικρό ποσοστό μόνο ελέγχεται από το δορυφόρο. Το επόμενο θέμα το αφορά την κατανομή των αλληλευτικών ποσοστώσεων. Τα κριτήρια για την κατανομή των ποσοστώσεων δεν ήταν πάντοτε ε, διαφανή. Ε, υπήρξε ένα πρόβλημα. Κάποια κράτη-μέλη ανέθεσαν την κατανομή των ποσοστώσεων στους οργανώσεις παραγωγών. Και υπήρξε πιθανό σύγκρουση, πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ενώ τα κριτήρια δεν ήταν πάντοτε διαφανή. Ε, έτσι, ε, συνιστούμε να ενημερώνεται η Κομισιόν για τα συστήματα κατανομής των ποσοστώσεων έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια και επίσης ε, προτείνουμε τη χρήση εναλλακτικών συστημάτων εντοπισμού για τα μικρά σκάφη. Το επόμενο θέμα αφορά τα δεδομένα της αλίας, τα οποία ήταν ανεπαρκή, ε, ε, ε, δεν ήταν πλήρη και ήταν αναξιόπιστα. Αυτό κυρίως όσον αφορά τα μικρά σκάφη που υποβάλλουν δηλώσεις σε χαρτί. Συνιστούμε την βελτίωση της επαλήθευσης των δεδομένων, κυρίως για τα μικρά σκάφη. Αυτό αφορά τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την Κομισιόν, η σύσταση είναι η δημιουργία και η, η, μιας πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών πληροφοριών για τα κράτη-μέλη και η προώθηση της, των, συστημάτων ηλεκτρονικής δήλωσης για τα μικρά σκάφη. Το τέλος, τελευταίο θέμα είναι τα συστήματα ε, ελέγχου. Ε, είναι λειτουργικά, όμως οι κυρώσεις δεν είναι πάντοτε αποτρεπτικές και εφαρμόζονται διαφορετικά. Δηλαδή δεν εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των, των αλλιέων. Συνιστούμε λοιπόν να επιβληθούν αποτρεπτικές κυρώσεις, κυρίως για τους ε, υπότροπους. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ε, παραβάτες που τιμωρούνται πέντε φορές το χρόνο και συνεχίζουν την πρακτική αυτή, που, πράγμα που δείχνει ότι το σύστημα κυρώσεων δεν είναι αποτελεσματικό. Η επόμενη σύσταση είναι πλήρης εφαρμογή ενός ε, συστήματος μορίων, ενός ποινολογίου, και ε, η πρόταση ενό συστήματος ανταλλαγής δεδομένων για τις παραβιάσεις και τις ε, κυρώσεις. Αυτά αφορούν την Κομισιόν. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τις ε, συστάσεις μας με θετικό πνεύμα και δήλωσε ότι θα τις εφαρμόσει συνεργαστήκαμε καλά με την Κομισιόν στη διάρκεια αυτού του ελέγχου και στη διάρκεια της διαδικασίας ε, αντιπαράθεσης. Ελπίζουμε ότι ο έλεγχός μας θα έχει θετικό αποτέλεσμα και θα οδηγήσει στη βελτίωση του συστήματος ελέγχου της Αλίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και με το λόγο στην Επιτροπή για τρία λεπτά. Καλημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Η Επιτροπή πραγματικά θεωρεί πολύ ευπρόσδεκτη την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση, διότι ε, το καθεστώς ελέγχου της Αλίας είναι πολύ σημαντικό σημαντικό για την αποτελεσματική εφαρμογή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και επειδή όμως φτάνει σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, ένα διάστημα όπου πρόσφατα η ίδια η Κομισιόν ολοκλήρωσε τη δική της αξιολόγηση του ε, κανονισμού ελέγχου. Χαιρόμαστε που τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου συνάδουν με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Κομισιόν. Θεωρούμε ότι παραμένουν σοβαρά προσκόμματα, ελλείμματα στον τομέα, στους τομείς που έχουν επισημάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Η εφαρμογή εκ μέρου των κρατών μελών δεν, είναι, ε, δεν γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο και δεν είναι απολύτως ικανοποιητική. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε τα κράτη-μέλη για την βελτίωση τη υλοποίηση και πρέπει να πω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει την, την υλοποίηση κάποιων από αυτές τις συστάσεις. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που θέτει το δικαστήριο αφορά το γεγονός ότι κάποιες διατάξεις του, ελέγχου, του κανονισμού ελέγχου πρέπει να τροποποιηθούν. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει με ικανοποίηση να ανακοινώσω, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα και στην Επιτροπή Ελίας, ότι η Επιτροπή πρόσφατα ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την ε, αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλίας. Δεν μπορούμε φυσικά να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα. Ε, μπορώ να σας, εξασφαλ... να σας διαβεβαιώσω όμως ότι θα λάβουμε στην πορεία υπόψη μας τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Εν γέννη λοιπόν συμφωνούμε απόλυτα, έχουμε ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή και όσον αφορά την αναθεώρηση του ε, κανονισμού ελέγχου θα λάβουμε υπόψη μας όλες τις τάσεις που έχουν γίνει. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστούμε πολύ. Πώς και δεν είχαν γίνει αυτά νωρίτερα, γιατί νομίζω ήταν αρμόδια η Επιτροπή να το ολοκληρώσει. Γιατί δεν έχει γίνει ήδη εδώ και καιρό αυτό. Αν ε, μπορείτε να μου απαντήσετε παρακαλώ σε αυτή τη συμπληρωματική ερώτηση. Yes. Ε, well, as I already said... Όπως σας είπα ήδη, η Επιτροπή πρόσφατα έκανε μία αξιολόγηση της υλοποίησης και του κανονισμού ελέγχου για να κρίνει αν είναι κατάλληλος. Όσον αφορά το επίπεδο υλοποίησης, η Επιτροπή κατέληξε, όπως και το ελεγκτικό συνέδριο, ότι είναι ανομοιόμορφο το επίπεδο υλοποίησης στα κράτη-μέλη και σε αρκετούς τομείς δεν είναι ικανοποιητικό. Ένας από τους τομείς όπου υπάρχουν οι περισσότερες ανησυχίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η επιβολή κυρώσεων. Είναι σημαντικό να επιβάλλονται κυρώσεις με ομοιόμορφο τρόπο, να είναι αναλογικές και αποτρεπτικές, διαφορετικά ε, πλήττεται η ίση μεταχείριση των αλλιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πρωτοβουλία επισκόπησης της κατάστασης σε όλα τα κράτη-μέλη και ίσως το μέλλον καταλήξει σε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις. Όσον αφορά την υλοποίηση, εντοπίστηκαν κάποια θέματα για την ε, υλοποίηση, μάλλον για την ε, μεταβίβαση δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων, καθώς και τη συλλογή δεδομένων. Ε, για τα δεδομένα για τα αλλιεύματα εντοπίστηκαν κάποιες ελλείψεις, αλλά αυτό το θέμα έχει πολλαπλές διαστάσεις. Έχει σχέση και με τον κανονισμό της υλοποίησης και για το, τη μελλοντική εκδοχή του κανονισμού και το ελεγκτικό συνέδριο επεσήμανε ότι υπάρχουν ακόμη κενά για τα δεδομένα σχετικά με τα ελιεύματα από ε, τους ε, μικρούς στόλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί και στην πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε πρόσφατα για την αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου, θα επικεντρωθούμε συγκεκριμένα στο σημείο αυτό. Υπάρχουν και πολλές άλλες παράμετροι, αλλά δεν έχουμε το χρόνο σήμερα για να διατρέξουμε όλες τις συστάσεις του Ελληνικού Συνεδρίου και όλα τα συμπεράσματα και όλες τις πιθανές δράσεις που θα λάβουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Δεν είναι εδώ εισηγητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα διανύμουμε το έγγραφο εργασία. Και περνάμε στο επόμενο σημείο τη μείσης διάταξη, που είναι η ειδική έκθεση 9 του 2017, στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία. Η κυρία Γιάκοψεν είναι υπεύθυνη για την παρουσίαση και σας δίνω το λόγο για την παρουσίαση της έκθεσης, κυρία Γιάκοψεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση για την καταπολέμηση της, ε, ε, της ε, εμπορίας ανθρώπων στην Νότια και Ανατολική Ασία. Ε, αυτό αποτελεί μια σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παγκόσμια απειλή κατά της ασφάλειας. Συνεπάγεται την ε, μεταφορά ανθρώπων δια της βίας ή με εξαπάτηση με σκοπό την εκμετάλλευση. Τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και κορίτσια και η πιο συνήθις μορφή εκμετάλλευσης είναι η καταναγκαστική εργασία και η σεξουαλική εκμετάλλευση. Όταν μιλάμε για ανθρώπινη, παράνομη διακίνηση ανθρώπων όλοι έχουμε διαφορετική εικόνα της κατάστασης κατάσταση. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία. Η, το, η Europol εκτιμά ότι ε, τα έσοδα από την παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι άνω των 29 ε, δις ευρώ. Επίσης εκτιμάται ότι περίπου 46 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε συνθήκες σύγχρονης ε, σκλαβιά, τα δύο τρίτα από αυτούς προέρχονται από την Ασία. Επίσης αξιολογήθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα έργων σε 10 διαφορετικές χώρες με σύνολο 31 εκατομμύρια ευρώ η καταπολέμηση της ε, παράνομη διακίνησης ανθρώπων είναι μακρόπνοη προσπάθεια και πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αίτια της παράνομη διακίνησης που είναι η ανισότητα των φύλων, η φτώχεια, η έλλειψη μόρφωσης και θέματα υγείας. Όσοι από εμά ε, απολαμβάνουμε χρόνο στους κήπους μας ξέρουμε ότι το ότι ε, πρέπει κανείς ε, να ε, έχει κανείς καλύτερα αποτελέσματα βγάζει τα ζυζάνια και τα εκριζώνει. Κατά την ίδια, με την ίδια αποτελεσματικότητα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες των ανθρώπων που, που, που πλήττουν τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Γι' αυτό αποφασίστηκε να επικεντρώσουμε τον έλεγχο σε, κάποια, σε κάποιες από τις χώρες προέλευσης αυτής της παρανομής διακίνησης. Μελετήσαμε τις περιοχές της Νότια και Ανατολικής Ασίας όπου επιμένει η παράνομη διακίνηση ανθρώπων και έχει αναγνωριστεί ως σοβαρό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό αποτελεί μια από τις προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Θέλουμε να εξετάσουμε αν η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης της περιοχές αυτές ήταν αποτελεσματική. Θέλαμε να δούμε αν είναι ολοκληρωμένη η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και αν τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά για την καταπολέμηση τη παράνομη εκείνη ανθρώπων στι περιοχέ αυτέ. Τι διαπιστώσαμε. Εν γέννη καταλήξαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέρη ήταν αποτελεσματική στην στήριξη της ε, ε, προσπάθεια για την καταπολέμηση τη παράνομης διακίνησης ανθρώπων στην περιοχή το πλαίσιο περιοχής, ε, το πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων εν μέρει είναι αποτελεσματικό. Όμως η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση εμπορίας δεν περιλαμβάνει στόχους ή συγκεκριμένους σκοπούς και αυτό θα βοηθούσε στις προσπάθειες επιτόπου και θα μπορούσε να βοηθήσει στο αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Διαπιστώσαμε ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπήρξε ιδιαίτερος χρήσιμο εργαλείο. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πετύχει την δημιουργία ειδικών εταιρικών σχέσεων για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων στην συγκεκριμένη περιοχή. Ένα άλλο μέσο που χρησιμοποιεί η Κομισιόν στην καταπολέμηση εμπορία εμπορίας ανθρώπων είναι η χρηματοδότηση διαφόρων έργων. Τα έργα αυτά πολύ συχνά ε, υλοποιούνται από τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διαπιστώσαμε ότι παρά τις αδυναμίες όλα τα έργα που μελετήσαμε έχουν δώσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Όμως η επίπτωση αυτού του αποτελέσματος θα μπορούσε να έχει μεγεθυνθεί και σε κάποιες περιπτώσεις το θέμα που μας απασχόλησε ήταν η βιωσιμότητά τους. Ενώ βλέπουμε γενικά βελτίωση την καταπολέμηση εμπορία ανθρώπων στην περιοχή, δύσκολα μπορούμε να συνδέσουμε αυτό την εξέλιξη στι συγκεκριμένε δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για την, από την κατανομή των πόρων, όσο και από τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Ο έλεγχο οδήγησε σε δύο γενικέ συστάσει. Γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν πρόκειται να υποβάλει μια νέα στρατηγική, ένα πλαίσιο πολιτική για την περίοδο μετά το 2016. Επίση, περιμένουμε να ε, δημοσιεύσει η Κομισιόν μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μέχρι τούδε αποτελεσμάτων μέχρι, ε, για την στρατηγική 2012-2016. Συνιστούμε λοιπόν στην ε, Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την στρατηγική για την ε, καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων ειδικά για την περιοχή και δεύτερον να βελτιστοποιήσει τις επιπτώσεις των έργων με το να το ενσωματώσει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Θα πρέπει να σκοπεύει στη στήριξη των έργων που περισσότερο θα συνεισφέρουν στην βιώσιμη καταπολέμηση τη εμπορίας ανθρώπων και να συνεισφέρει περισσότερο στην συνεργασία και τι συνέργειε μεταξύ των έργων. Η αντιμετώπιση της παράνομης εμπορία ανθρώπων απαιτεί συνέργειε και συνεχή ε, δράση. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρου τη Γενική τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση αυτή. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει για την αντιμετώπιση Τη εμπορία ανθρώπων στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία. Συμφωνούμε ότι η καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων στην περιφέρεια αυτή έχει συνολικά βελτιωθεί, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσει η καλή προσπάθεια. Η ε, Επιτροπή θεωρεί ε, το θέμα της καταπολέμησης ε, της εμπορίας ανθρώπων ε, να πω στο κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές και σε θέματα ασφάλειας. Γίνεται όλο και περισσότερο επικοδομητικό διάλογο με χώρε τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία για το θέμα, σε περιφερειακέ μορφέ και σε βήματα όπω η ΑΣΕΑΝ και η ΑΣΕΜ καθώς και σε ευρύτερα βήματα για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πόρους, καθώς ε, και εντατική συνεργασία με κάθε συμβαλόμενο. Καταγράφουμε τα επιτεύγματά μας ε, και την διαδικασία που ακολουθούμε με την παρούσα στρατηγική. Εξετάζουμε τις τάσεις, τα προβλήματα, αξιολογούμε, συζητούμε με όλους τους εμπλεκομένους στις μελλοντικέ δράσεις που ίσως χρειαστούν. Ο κύριος στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που θέτει μέσω συντονισμού και μέσω μιας συνεκτικής προσέγγισης, ούτως ώστε να έχουμε ε, συγκεκριμένε λύσει βάσει των αναγκών, όπω συνιστά και το ελεγκτικό συνέδριο. Πιο συγκεκριμένα για τι συστάσει του ελεγκτικού συνεδρίου, όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του στρατηγικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να εφαρμόσει αυτή τη σύσταση, ιδίω μέσω ενό ε, νέου καταλόγου προτεραιοτήτων που σκεφτόμαστε να προτείνουμε για τι ε, πολιτικέ που θα ακολουθήσουμε μετά το 2016 για την εμπορία ανθρώπων θα συνεχίσει να παραμείνει ε, στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας ε, κατά το διάλογο με τις ε, εμπλεκόμενες χώρες. Θα χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα τα οποία έχουμε αποκομίσει από προηγούμενες δράσεις και σχετικά έγγραφα και θα δοθεί και επιχειρησιακή καθοδήγηση για τις δράσεις επιτόπου. Θα επεκταθούν σχετικές οδηγίες και θα υποβάλλονται αντίστοιχες εκθέσεις. Όσον αφορά τη δεύτερη σύσταση, το, τα έργα που ανέλησε το ελεγκτικό συνέδριο υλοποιήθηκαν σε δύσκολα περιβάλλοντα από πλευρά πολιτικής. Η βιωσιμότητα των έργων πάντοτε είναι σημαντική για την Επιτροπή και για τις αντιπροσωπείε των κρατών μελών. Για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα κάποιων δράσεων, όπως η άμεση βοήθεια στα θύματα, ε, οι προκλήσει είναι πολλαπλέ. Βεβαίως, στο μέλλον θα εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας στα θέματα τα οποία επισημαίνει το ελεγκτικό συνέδριο για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων στις πιθανές χώρες προτεραιότητας στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία. Ο κ. Σελαφράγκα είναι ο εισηγητή μα, σα δίνω το λόγο. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις εισηγήσεις ε, που ε, ακούσαμε σήμερα για αυτό το φρικτό θέμα, το εμπόριο ανθρώπων όπου σχεδόν το 80% είναι γυναίκες, αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ε, είναι θύματα γάμων με ανήλικα, ε, είναι πραγματικά κάτι στο οποίο θα πρέπει άμεσα να ενεργήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή το σημασία που, την έκταση που παίρνει αυτό το φαινόμενο. Μιλάμε για 40 και βάλε εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάμε για νούμερα εγκληματικότητας μεγαλύτερα από αυτά του εμπορίου όπλων και θα πρέπει να δούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πληγή. Ακούσαμε ότι τα έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέχρι στιγμής μερικώς αποτελεσματικά και αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί αυτό το φαινόμενο είναι, έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και εμείς θέλουμε να παίξουμε το ρόλο στρατηγικού εταίρου για τις χώρες της ε, Ασίας όπως είδαμε και με τις τελευταίες συμφωνίες με την Ταϊλάνδη, την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε αυτή την προτεραιότητα που είναι σύμμορφη προς τις ε, αξίες και τις αρχές που εμείς υπερασπιζόμαστε. Λαμβάνουμε υπόψη και σημειώνουμε με μεγάλο ενδιαφέρον επίσης Πρόεδρε τις παρατηρήσεις και τις αντιδράσεις της Κομισιόν ενώπιον αυτού του προβλήματος που πρέπει να λυθεί μέσω συνεργασίας της Επιτροπής της ΕΙΕΔ και των δημοσιονομικών μέσων που έχουμε, δηλαδή αναπτυξιακή βοήθεια, ανθρώπινα δικαιώματα και ε, πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και σημείωσα με, θετικό, με θετική μνήμα τη διαθεσιμότητα της Κομισιόν για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, δηλαδή να δούμε πώς θα τοποθετήσουμε σε πιο στρατηγικό πλαίσιο τη δράση μας και επίσης πώς θα μπορέσουμε να μάθουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος ότι δηλαδή ναι, τα στοιχεία είναι καλύτερα, αλλά αυτό το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο, αν τελικά οφείλονται στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν οφείλονται σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει οι δράση μας θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, πιο ε, συνεχτική, πιο ολοκληρωμένη και μέσα από τους εθνείς οργανισμούς όπως ο ΙΕ, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να καλέσω την Κομισιόν όντως σε, σε αυτό το δρόμο που έχει χαράξει να λάβει υπόψη αυτές τις ε, προτάσεις για να δούμε πώς θα μπορέσουμε όλοι να κάνουμε κάτι καλύτερο με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας από τα δημοσιονομικά μας μέσα, ώστε να φτάσουμε σε πιο αποτελεσματικές δράσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλο κομμάτι αυτού, α, μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων φτάνει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. 200 με 400 χιλιάδες θύματα από όλα αυτά τα εκατομμύρια έρχονται, φτάνουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μπορέσουμε λοιπόν με τις περιφερειακές και τις διμερείς συμφωνίες που έχουμε να πρέπει να <clears throat> βρούμε με τους συνομιλητές μας κάποιο διάβλο που θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον προγραμματισμό ε, και στον αγώνα κατά αυτού ε, του, αυτής της ντροπής όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει απάντηση και να είναι πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε και αυτό το σημείο της ημερησία διάταξης. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Τσέλε που είναι ο εισηγητή ε, τη προηγούμενη έκθεση για την Αλία και δεν ήταν παρόν προηγουμένω. Ευχαριστώ. Ε, πιο πολύ ώρα έκανα να έρθω από το αεροδρόμιο στο Κοινοβούλιο παρά από το Βερολίνο στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ποσισόσκη και την ομάδα του εκ μέρους του ε, ελεκτικού συνεδρίου. Αφιέρωσαν πολύ χρόνο και προσπάθεια για την έκθεση αυτή για την αλία. Δεν είναι ε, ικανοποιητική η κατάσταση είχαμε συμφωνήσει διάφορα θέματα για την βιώσιμη αλληλεία και για τα αλληλευτικά αποθέματα, ούτως ώστε να υπάρχουν αλληλευτικοί πόροι και για τις ε, επόμενες γενναίες, αλλά τα κράτη-μέλη παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις στο κατά πόσο υλοποιούν όλα αυτά. Και γι' αυτό υπάρχουν ε, και παράπονα και καταγγελίες εκ μέρους ε, των πολιτών, εκ μέρους των αλλιέων όταν υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι κανόνες, ε, θα πρέπει οι κανόνες αυτοί ε, να εφαρμόζονται στην πράξη, να υλοποιούνται τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, αλλά εδώ βλέπουμε ότι γίνονται στα κρυφά αυτά τα οποία γίνονται, δεν τηρούνται οι κανόνες, ε, κάποιοι ε, παραβαίνουν τις διατάξεις και νομίζω ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου θα αποτελέσει μια καλή βάση για να μπορέσουμε εκ νέου να επισημάνουμε τα προβλήματα σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ακρόαση για το θέμα αυτό τώρα μάλιστα που έχουμε σαν βάση την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και μπορούμε σε συνεργασία με φορείς από τον τομέα της αλληλείας να οργανώσουμε μια τέτοια ακρόαση και να καλύψουμε θέματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο. Σας ευχαριστώ πολύ που με επιτρέψατε να λάβω το λόγο καθυστερημένο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος δίνουμε 10 λεπτά σε κάθε έκθεση και βέβαια δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ε, για να ασχοληθούμε ε, ενδελεχώς με κάθε θέμα. Υπάρχει λοιπόν αντικείμενο και θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ακρόαση για να συζητήσουμε τα θέματα της Ελίας λεπτομερέστερα. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Είναι η έκθεση υπαριθμών 10 του 2017, στήριξη προς τους νέους γεωργούς ούτως ώστε να είναι καλύτερη προώθηση της αποτελεσματικής ανανέωσης των γενεών. Οι εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου καλό είναι να χρησιμοποιούνται ε, ως βάση και εδώ μπορούμε να δούμε ε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ανανέωση ε, των ασχολημένων με τη γεωργία. Θα δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Βογεσόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με το αν θα πρέπει να γίνει καλύτερη στόχευση στις ενισχύσεις που καταβάλλονται στους νέους γεωργούς. Ε, μπορώ να χρησιμοποιήσω και την παρουσίαση αυτή τη φορά. Θέλω να σας ενθαρρύνω να μελετήσετε τα δεδομένα αυτά της έκθεσης, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα πρέπει να μας ανησυχήσουν. Δείχνουν ότι ο πληθυσμός των ε, γεωργών την τελευταία δεκαετία από το 2005 μέχρι το 2013 μειώθηκε από 14,5 εκατομμύρια σε 10,7 εκατομμύρια. Χάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 4 εκατομμύρια αγροκτήματα, ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις τη δεκαετία πάνω από 30.000 ε, αγροκτήματα το μήνα και πάνω από χίλια αγροκτήματα την ημέρα. Και βεβαίως όσον αφορά τους νέους γεωργούς, ο πληθυσμός τους δυστυχώς μειώθηκε από 3,3 εκατομμύρια το 2005 σε 2,3 εκατομμύρια το 2013. Και στο, στη διαφάνεια αυτή, στο σχεδιάγραμμα αυτό βλέπουμε τη μείωση του πληθυσμού των γεωργών, όπως επίσης και οι εκτάσεις που κατέχουν μειώθηκαν από 58 εκατομμύρια εκτάρια σε 52 εκατομμύρια εκτάρια. Ο πληθυσμός μειώθηκε, αλλά και οι εκτάσεις που κατέχουν οι νέοι ε, γεωργοί μειώθηκαν. Θεωρώ ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι το εξής. Μόνο δύο κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθυσμός των νεότερων γεωργών κάτω των 35 ετών είναι άνω του 10%. Η Αυστρία και η Πολωνία είναι αυτά τα κράτη-μέλη. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τρία μόνο κράτη-μέλη στα οποία ο πληθυσμός των πιο ηλικιωμένων ε, αγροτών άνω των 65 είναι κάτω του 10%. Μάλλον το ποσοστό, όχι ο πληθυσμός. Το ποσοστό αυτών των αγροτών είναι κάτω του 10% μόνο στη, σε τρία κράτη-μέλη, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία. Στην Πορτογαλία όμως ο πληθυσμός των άνω των 65 ετών είναι πάνω από 50%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανούμε περίπου 10 δις ευρώ για την στήριξη των νέων γεωργών στην ε, περίοδο μέχρι το 2020 και δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η δαπάνη αυτή έχει θετική, ε, θετικό αποτέλεσμα τουλάχιστον στην ανανέωση της, των γενεών. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει ανανέωση των γενεών, αλλά εν γέννη δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσής μας είναι... Πρέπει Μάλλον υπάρχουν ελάχιστε ενδείξει ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη έχει διευκολύνει την εγκατάσταση νέων αγροτών και έχει βελτιώσει την ανανέωση των γενεών. Συνιστούμε να βελτιώσουν την παρακολούθηση, ούτω ώστε να συγκεντρώνονται δεδομένα που αφορούν το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Είναι η γέννη εν γέννη ανάγκες των νέων ε, γεωργών δεν αναλύθηκαν επαρκώς και μόνο εν μέρη ε, καλύπτονται οι ανάγκες τους από το υπάρχον πρόγραμμα. Ζητάμε να βελτιωθεί η λογική της παρέμβασης με μια σωστή αξιολόγηση και καθορισμό των ε, στοιχείων της. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα κράτη-μέλη. Δεν είναι πρόβλημα περιφερειών οι γεωργών. Δεν βρήκαμε καταχρήσεις εκ μέρους των αγροτών. Το πρόβλημα βρίσκεται στην ίδια τη λογική της παρέμβασης η οποία δεν είναι σωστή. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας. Ενδεχομένως το πρόβλημα να βρίσκεται στο ότι προσπαθούμε να ε, ε, αντιμετωπίσουμε διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικές καταστροφές ε, στην Ευρώπη με το ίδιο φάρμακο. Γιατί η κατάσταση διαφέρει, η ηλικιακή δομή διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Κάποια είναι σε καλύτερη κατάσταση, κάποια άλλα... Ας πούμε, υπάρχουν κράτη-μέλη που ο πληθυσμός άνω των 65 ετών είναι κάτω από 10%, ενώ σε άλλα είναι 50%. Το μέλλον της ΚΑΠ θα πρέπει να στοχευθεί καλύτερα όσον αφορά τα συγκεκριμένα προβλήματα κάθε κράτους μέλους. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την δυνατότητα να παρουσιάσω την έκθεση, η οποία ελπίζω ότι θα βοηθήσει τη μελλοντική τη συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ. Σας ευχαριστούμε ανησυχητικά τα στοιχεία. Θα δώσω ε, στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας το λόγο, κύριε Λουίς Χόφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη τη Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει αυτή την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συμφωνούμε με την άποψη του Ελεκτικού συνεδρίου ότι είναι ζωτική σημασία η στήριξη προ του νέου αγρότε, για να μπορέσει η γεωργία να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα και για τι μελλοντικέ γενιές και κατά την προετοιμασία τη νέα περίοδου το έχουμε σκεφτεί και βελτιώσαμε τα εφιστάμενα μέτρα στο δεύτερο πυλώνα και προσθέσαμε ένα επιπλέον στοιχείο ένα επιπλέον στοιχείο στήριξης της άμεσης ενισχύσης. Θα ήθελα τώρα να επισημάνω κάποια σημεία της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Το πρώτο είναι το πεδίο του ελέγχου. Έχουμε δύο διακεκριμένα συστήματα στήριξης. Στον πρώτο πυλώνα αυτό που κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε ε, τα οικονομικά προβλήματα κατά τα πρώτα έτη εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση. Και ο νέος αγρότης λαμβάνει μια επιπλέον πληρωμή πέραν των άμεσων ενισχύσεων, μια πρόσθετη λοιπόν στήριξη για να ληφθεί υπόψη η δική του κατάσταση. Αυτό είναι υποχρεωτικό στοιχείο που πρέπει όλα τα κρατη να το εφαρμόζουν. Το ελεγκτικό συνέδριο στην ανάλυση του λαμβάνει υπόψη μόνο αυτή την πρόσθετη πληρωμή που δίδεται στους ε, νέους αγρότες που είναι 2,6 δισεκατομμύρια σε όλη την περίοδο αυτό το ποσό είναι μικρότερο σε σχέση με τη συνολική προσπάθεια που καταβάλουμε κατά την περίοδο 2015-2020. Ε, για τους νέους αγρότες καταβάλλονται 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες οικονομικές ανάγκες και αβεβαιότητα κατά την έναρξη δραστηριότητα, θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους γεωργούς και γι' αυτό χορηγούμε αυτά τα κονδύλια. Τώρα, ε, σύμφωνα με τον ε, ε, άλλο ε, πυλώνα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη λογική των νέων γεωργών αλλά με πιο συγκεκριμένη στήριξη. Δηλαδή, περιλαμβάνεται μια δέσμη μέτρων μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν τα κράτη-μέλη και να σχηματίσουν τη δική τους δέσμη μέτρων και να αποφασίσουν τι είδους στήριξη θέλουν να δίνουν στους νέους γεωργούς βάσει αξιολόγησης των αναγκών τους. Αλλά αυτή την αξιολόγηση πρέπει να την κάνουν τα κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε μια πλήρη συνταγή για επίλυση των προβλημάτων των αγροτών σε όλα τα κράτη-μέλη, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετική η κατάσταση από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ακριβώς αυτό είπε και το Ελληνικό Συνέδριο. Τα κράτη-μέλη επιλέγουν τα συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου και επιλέγουν στοχευμένα μέτρα καταγράφουμε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τους νέους αγρότες όσον αφορά τις επαγγελματικές τους ικανότητες για να μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Θα πρέπει να υποβάλουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να λάβουν τη στήριξη και υπάρχει στόχευση μέσω κριτηρίων επιλογής. Αυτό ήδη το θεσπίζει ο κανονισμός και τα κράτη-μέλη πρέπει να επιβάλλουν το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης για τη στήριξη των νέων αγροτών. Αυτά είναι κάποια στοιχεία λοιπόν ε, που σχηματίζουν το πακέτο στήριξης των νέων γεωργών. Σύμφωνα με το δεύτερο πυλώνα, το κονδύλι είναι 6,7 δισεκατομμύρια και θα στηριχθούν 177.000 νέοι γεωργοί σύμφωνα με τα στοιχεία των κρατών μελών. Κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δύο πυλώνες έχουν εξορισμού υποχρεωτική στήριξη, γιατί έτσι είναι δομημένο το πρόγραμμα. Υπάρχει μια επιπλέον δυσκολία που πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα μόνο με τους νέους γεωργούς, αλλά και με τους ε, ε, μεγαλύτερους ηλικία γεωργούς, οι οποίοι δεν εγκαταλείπουν την αγροτική εκμετάλλευση. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις και κρατούν την εκμετάλλευσή τους για να συνεχίσουν την επαγγελματική δραστηριότητα ε, ούτως ώστε να μην χάσουν τα δικαιώματα απασχόλησης τα οποία έχουν λόγω των δυσμενών συνθήκων σε πολλά κράτη-μέλη. Εδώ χρειάζεται μια επανεξέταση των μέτρων για την επόμενη περίοδο για να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έχουμε λάβει υπόψη τη σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου και έχουμε δεσμευθεί ότι θα το εξετάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για το τι ακριβώς θα κάνουμε κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τα κράτη-μέλη στον καλό σχεδιασμό των μέτρων στήριξης και στον προσδιορισμό των αναγκών που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος. Στόχος μας είναι να έχουμε καλύτερη στόχευση των μέτρων. Αυτό είναι αυτονόητο. Και χρειάζεται συνεργασία με τα κράτη-μέλη για την ε, κατάρτιση δικτών και αυτό είναι τμήμα της γενικότερης ε, πολιτικής που θα πρέπει να αποδίδει καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε πει να δώσουμε 10 λεπτά σε κάθε έκθεση, αλλά θα πρέπει να τηρείτε το χρόνο ομιλίας και μέχρι τώρα κανείς δεν έχει τηρήσει το χρόνο ομιλίας. Θα δώσω λόγο στη συνάδελφο Κάντενμπαχ. Μπορώ κι εγώ να μην τηρήσω το χρόνο ομιλίας. Η κυρία Γιάκοψεν ήταν η μόνη που τήρησε τον χρόνο της. Το συγγνώμη κυρία Γιάκοψεν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κάντενμπαχ. Ευχαριστούμε το ελεγκτικό συνέδριο και τον κύριο Βοτσεσόφσκι, πρώην συνάδελφο. Νομίζω ότι δείχνει με δραματικό τρόπο η έκθεση ότι δεν επιτυχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι βλέπουμε ότι δεν είναι επαρκείς οι νέοι αγρότες, δεν είναι επαρκείς η ε, ε, πρόοδηση των νέων αγροτών ώστε να μένουν ε, και να προωθούν τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου. και από την παρουσίαση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας είδαμε ότι δεν έχουν επιτευχθεί τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε όχι μόνο βιοπικιλότητα, αλλά χρειαζόμαστε και ε, διάφορες μορφές μέτρων ανάλογα με το είδος των εκμεταλλεύσεων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ειδών διατροφής στην Ευρώπη, την ασφάλεια της αλυσίδας διατροφής και αυτό μέσω της επιδίωξης των καλύτερων πρακτικών. Και χρειάζεται μια ε, συζήτηση από αυτού για να δούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα το επιτύχουν. Ακούσαμε αυτό που μας είπε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και βλέπουμε ότι ένα σύνολο μέτρων, δεν μιλάμε μόνο ε, για ένα ε, δίκτυο ασφαλείας, δίκτυο κοινωνικής ασφαλείας, μιλάμε και για την διάρθρωση της υπαίθρου και για την ε, περιφερειακή πολιτική διότι θα πρέπει να προσφέρουμε στους νέους ε, γεωργούς έναν χώρο που θα είναι ελκυστικό, ούτως ώστε να θέλουν να είναι σε ένα χώρο της υπαίθρου ή σε ένα ορεινό ε, περιβάλλον. Και μέσω του πολιετούς ε, προγράμματος μπορούμε να δούμε πώς να δώσουμε ένα τέτοιο χαρακτήρα στην κοινή γεωργική πολιτική, ούτως ώστε να προωθούμε τις πολιτικές ε, που επιθυμούμε, όχι μόνο ε, από πλευράς ε, ποσοτικών στόχων, αλλά και από πλευράς ποιοτικών στόχων και διαφοροποίησης. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή τη σύντομη παρουσίαση σήμερα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με ένα έγγραφο εργασίας στο οποίο θα καθορίζονται όλα αυτά τα θέματα και θα μας δώσει και την ευκαιρία να συζητήσουμε λεπτομερέστερα πώς μπορούμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία διαπιστώνουμε μετά από την παρουσίαση της σημερινής έκθεσης. Ίσως να χρειάζεται κάποιος ευέλικτος χαρακτήρας, ιδίως στο δεύτερο πυλώνα, για να μπορούμε να έχουμε και καλό υπολογισμό των επιτευγμάτων των μέτρων σε κάθε κράτος μέλος, γιατί βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, παρουσιάζουν αποτελέσματα με διαφορετικό τρόπο και δεν μπορούμε να ξέρουμε ε, ποιο είναι το επιθυμητό σύστημα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Προτείνω να βάλουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη άλλη μια φορά, με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένε ακροάσει ή συζητήσει ή έγγραφα τα οποία προτείνουμε για να έχουμε μια επαρκή παρακολούθηση. Δηλαδή όχι μόνο δεν επιτυχάνουμε το στόχο, αλλά παρεμποδίζεται και η επίτευξη του στόχου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να το επιλύσουμε. Πρέπει να σας πω ότι μόνο οι συντονιστέ αποφάσισαν ότι θα δίδεται ο λόγο μόνο στον εισηγητή κάθε θέματο. Οπότε δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε άλλου ομιλητέ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο που είναι η θέση μα για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και δίνω το λόγο στον συνάδελφο Σαβάμα. Επαναλαμβάνω στα αγγλικά για όσους δεν με άκουσαν ότι συμφώνησαν οι συντονιστές ότι θα δίνεται ο λόγος μόνο στον εισηγητή κάθε θέματος. Οπότε περνάμε στο επόμενο θέμα, θα 13 και το λόγο στον κύριο Σαρβάμα. Thank you, Madam Chair. Um, well, I will go straight. Ευχαριστώ. Εγώ θα περάσω αμέσω ε, στο θέμα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αναμένεται η να το δημοσιεύσει τον Ιούνιο του 2018 είτε το αργότερο του Σεπτέμβριο. Γι' αυτό και η ε, Επιτροπή Προπολογισμού προετοιμάζει έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ώστε να μπορέσει να, το Κοινοβούλιο να παρουσιάσει την άποψή της για το PDP και να επηρεάσει ελπίζουμε και την πρόταση, τη, ε, πρόταση της Επιτροπής εκ των προτέρων. Από ό,τι άκουσα η Κομισιόν ήδη προχωρεί και μάλιστα έχει προχωρήσει σε βάθος στην προετοιμασία. Εμείς, ε, ο, η Επιτροπή Προϋπολογισμού, Ελέγχου Προϋπολογισμού, θα είμαστε μια από τις επιτροπές που θα συμβάλλουμε με τη δική μας γνωμοδότηση. Δική μου αφεντηρία για αυτή την γνωμοδότηση είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη επιρροή γίνεται και στα θέματα τα δημοσιονομικά. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε πίσω, γιατί όπως ε, λένε και οι συγητές Όλμπριχτ και Θώμα της Επιτροπής Προπολογισμού, Σαφώ. η δική του πρωτοβουλία θα αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα αφορά τα δημοσιονομικά θέματα και το δεύτερο τμήμα θα αφορά τομεί πολιτικής επί τη βάση των νομοδοτήσεων των ε, επιμέρους επιτροπών. Και ήδη το έχω συζητήσει αυτό επί μακρόν με την Επιτροπή Προπολογισμού και πιστεύω πως έχουμε καλές πιθανότητες να προετοιμάσουμε εις βάθος και εκτεταμένη ε, γνωμοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν έχω κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σημεία μάλλον που θα ήθελα ήδη να τα σχολιάσετε όσοι ενδιαφέρεστε και να συμβάλλετε ήδη σε αυτό το πρώιμο στάδιο γιατί όσον αφορά το πρόγραμμα εγώ έχω ταυτόχρονα προσπαθήσει και έχω πιέσει όσο γίνεται περισσότερο του, τις προθεσμίες. Τώρα, ο προπολογισμό θα έχει το έτοιμο, το έτοιμο το κείμενό του το Δεκέμβριο και το πρόγραμμα του έχει έτσι ώστε να συζητήσουν τα θέματα την ίδια πρωτοβουλία μάλλον τον Ιανουάριο, να το ψηφίσουν στην Επιτροπή το Φεβρουάριο και ο στόχος είναι όλα να έχουν ετοιμαστεί για την Ολομέλεια του Μαρτίου. Εγώ θα προσπαθήσω να καθυστερήσω όσο γίνεται αυτή την ε, προθεσμία. Αυτό σημαίνει ότι τώρα εξετάζουμε αυτή το σχέδιο έκθεσης είτε στις 11 είτε στις 12 Οκτωβρίου. Με άλλα λόγια, το σχέδιο γνωμοδότησης μάλλον θα το έχετε στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, πράγμα που μας δίνει μια καλή ευκαιρία ε, να το σκεφτούμε στη διάρκεια των ε, θερινών διακοπών και θα τα πω σύντομα γιατί δεν θέλω να ε, σπαταλήσω το χρόνο μας, αλλά σύντομα σύντομα να σας δείξω τις, κάποιες από τις ιδέες που έχω μέσα στιγμής και φυσικά είναι ανοιχτά όλα αυτά σε συζήτηση. Αν δούμε τους τίτλους, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να έχουμε εμείς ε, γνώμη για διάφορα δημοσιονομικά θέματα και όχι μόνο για τον έλεγχο προπολογισμού. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν με τον έλεγχο προπολογισμού, η αναθεώρηση των δαπανών της Ένωσης είναι ένα από τα θέματα ε, τα οποία θα πρέπει να κάνει σωστά η Κομισιόν ώστε να μπορέσει μετά να προγραμματίσει για το PDP μετά το 2020. Θα πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε πολύ ξενυχιστική μελέτη των δαπανών ώστε να αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο η χορήγηση πόρων μέσα στον προπολογισμό αντικατοπτρίζει πραγματικά τις στατικικές μας προτεραιότητες. Επίσης με αυτό συμβαδίζει και το δημοσιονομικό θέμα των recitals. Έχουμε ήδη ένα ψήφισμα που ζητά να ε, προχωρήσουμε από τα 7 στα 5 χρόνια και νομίζω πως αυτό είναι ένα καλό σημείο κίνησης για καλύτερο προγραμματισμό. Τώρα, τα απορίσματα αυτής της ε, μελέτης των δαπανών θα μας επιτρέψουν να ε, ε, να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τα χρήματα και επίσης πώς ε, και κατά πόσον είναι αξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει να προσέξουμε περισσότερα είναι το πώς συμβαίνουν οι απάτες και πώς μπορούμε να τις προλάβουμε και οι παρατυπίες. Και η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει να είναι μέσα στο ίδιο καλάθι. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλο ένα και περισσότερο πώς θα εστιάσουμε σωστότερα τους πόρους του, του ελέγχου, ώστε να μας όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. στόχοι και προτεραιότητες. Ευελιξία. Ο προϋπολογισμός οφείλει να προσαρμόζεται σε απρόσμενες αλλαγές και περιστάσεις. Οπότε είναι και αυτό για εμάς ενδιαφέρον να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι ό,τι κάνουν στο προγραμματισμό του PDP θα έχει νόημα και τα επόμενα χρόνια όταν θα κοιτάξουμε αναδρομικά τι συνέβη. Θα πρέπει επίσης να ζητήσουμε και άλλη απλοποίηση και λιγότερο γραφειοκρατικό φόρτο. Θα μπορούσαμε λοιπόν όλα αυτά να τα βάλουμε στο, στη γνωμοδότησή μας. Επίσης, κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες ε, γραμμές ε, για τον προϋπολογισμό επί τη βάση επιδόσεων, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ιεράρχηση στόχων και να ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Να μην μπούμε βέβαια στις δικές σας, στις, στους ορισμούς, γιατί δεν είναι αυτό δικιά μας δουλειά αλλά γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία ώστε να δώσουμε τις ιδέες μας για το πώς θα μπουν χρήματα καταρχάς στον προπολογισμό μετά το Brexit. Πώς θα καλυφθεί το κενό του Brexit. Το κενό που θα αφήσει πίσω του το Brexit. Θα είναι κάτι που θέλω να συμπεριληφθεί Έχω κάποιες πρωταρχικές ε, σκέψεις, αλλά ίσως είναι πολύ νωρίς για να μπούμε σε τέτοια λεπτομέρεια, εκτός ε, αν βεβαίως σας ενδιαφέρει και θέλετε να το συζητήσουμε. Τα... Είναι αυτό επαρκές για την ανταλλαγή απόψεων τη σημερινή. Να Νομίζω πως τελικά πριν να έχουμε το σχέδιο να σας πω ότι το πρόβλημα που έχω είναι πώς θα ορίσουμε το πεδίο εφαρμογής, το εύρος μάλλον, ώστε να έχουμε μια <clears throat> σύντομη και περιληπτική γνωμοδότηση χωρίς να υπερβάλλουμε. Αυτά, Πρόεδρε, αυτά έχω για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Άλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Σαββάμα. Θα ήθελα και εγώ να πω την γνώμη μου για το τι μπορούμε να κάνουμε με το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα να προτείνω να εξετάσουμε την εικόνα γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τον ετήσιο προπολογισμό που εκπονείται κάθε χρόνο και υπάρχει το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι περίοδο 5 7 έτη. Α υποθέσουμε ότι από την επόμενη φορά η διάρκεια θα είναι πενταετή. Θα έχουμε λοιπόν ένα πενταετέ πρόγραμμα και ένα ετήσιο προπολογισμό. Κάτι λείπει στην ευρύτερη αυτή εικόνα. Πού βρίσκεται η μακροπρόθεσμη εικόνα δεκαετής, δεκαπενταετής διάρκεια. Το ετήσιο πρόγραμμα έχει λεπτομερείς ε, οικονομικές προτάσεις. Το πολιτεύθυνο οικονομικό πλαίσιο είναι μεσοπρόθεσμο και μας λείπει το μακροπρόθεσμο που είναι η δήλωση των προθέσεών μας. Για να είμαστε αποτελεσματικοί ε, και να επιτύχουμε προστιθέμενη αξία για την κατανομή των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη εικόνα για το τι θα συμβαίνει τουλάχιστον 10 χρόνια από τώρα. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα θέλουμε να επιτύχουμε σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία. Είχαμε τη στρατηγική του 2020, τώρα θα χρειαζόμαστε μια στρατηγική 2030 και να υπάρχει παράλληλα και ο μεσοπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός. Κάτι ακόμη τώρα. Όσον αφορά τις ε, πληρωμές, θα θυμάστε τη συζήτηση στο τέλος του 2014 για τα υπόλοιπα προς εκαθάριση. Μπορούμε να διδαχθούμε λοιπόν για το πώς πρέπει να κάνουμε τη διαχείριση του προϋπολογισμού στο μέλλον για να μην προκύψει πάλι μια τέτοια ε, δύσκολη κατάσταση. Στο τωρινό σύστημα εκπονούνται τα συστατικά του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μια φορά κάθε 7 χρόνια και στο μέλλον μια φορά κάθε 5 χρόνια. Μετά τελειώνουν απότομα και ξεκινάνε όλα από την αρχή για το επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Για να αποφύγουμε τέτοιου είδους μειονεκτήματα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κυλιόμενο σύστημα για αυτά τα πλαίσια. Κάθε πολιετές λοιπόν δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχει παρόμοια διάρκεια με το επόμενο, αλλά το επόμενο πολιετές πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει εν μέρη και το προηγούμενο. Να υπάρχει λοιπόν μια επικάλυψη χρονική, ούτω ώστε να αποφεύγονται οι εχμές και τα χαμηλά σημεία στην αρχή και στο τέλος κάθε πολιετούς πλαισίου. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντε, δύο λεπτά. Ο κύριος Πρώτα ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να συγχαρώ τον Πέτρη Σαββάμα για την παρουσίασή του. Ήταν πολύ ισορροπημένη και ε, κατάλληλη για την ε, τωρινή μας κατάσταση. Ο Πέτρη μας ε, παρουσίασε τα πιο κέρια σημεία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Ε, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να έχουμε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση πόρων. Να κάνουμε συστάσεις για προγραμματισμό στους τομείς όπου θα έχουμε τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική η οποία μόλις εγκρίθηκε στη δήλωση της Ρώμης το Μάρτιο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 για μας θα είναι πολύ σημαντικό το θέμα του Brexit στη συνέχεια, διότι μετά το Brexit ε, το μέσο κατακεφαλήν ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Το χαμηλότερο λοιπόν κατακεφαλήν ΑΕΠ ως μέσος όρος θα επηρεάσει και την πολιτική συνοχής και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα αλλάξει η κατανομή πόρων στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είτε επταετές είτε πενταετές, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Σημαντικό είναι τι επιπτώσεις θα υπάρξουν. Και έχουμε και διακηρύξεις για την Ευρωζώνη που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά συνεχίζεται η συζήτηση. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Όπως πολύ σωστά είπε ο Πέτρη, θα πρέπει να περιμένουμε προς το παρόν και να δούμε τι θα υποβληθεί για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε εγκαίρως. Θέλουμε να συνεισφέρουμε ώστε να έχουμε ένα καλύτερο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο από ό,τι τα προηγούμενα. με τις απαραίτητες απλουστεύσεις και με τη μείωση του περιθώριου σφάλματος, όπως είπε ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη γιατί έχω μια άλλη συνάντηση στην οποία πρέπει να πάω και θα χρειαστεί να φύγω. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μέχρι τώρα. Η κυρία Γιάννα Ζέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαραβάμα και αυτή, για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Θα ήθελα να θυμίσω στην, ε, καταρχάς ότι το ελεγκτικό συνέδριο και νομίζω ε, ήταν ε, ο κύριος Ήταλα μας θύμισε ότι είναι τμήμα των σφαλμάτων το γεγονός ότι δεν δίνεται τα απαραίτητα κονδύλια μέσω του προπολογισμού στα προγράμματα και στα έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί και προβλέπονται. Χρειάζεται λοιπόν από την Κόντο να μπούμε στο σχεδιασμό, να παρέμβουμε στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού, του PDP, στο σχεδιασμό των ίδιων πόρων, ώστε να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τις φιλοδοξίες, τα προγράμματα, τα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτά να τα συσχετίσουμε ε, με τους πόρους που όλο ένα και μειώνονται. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη και να το λύσουμε. Με ποιο τρόπο δηλαδή θα μπορέσουμε να καλύψουμε και το πρόβλημα του Brexit με περισσότερους ίδιους πόρους ή καλύτερους ίδιους πόρους. Σε αυτό το PDP που ονομάζεται μετά το 2020 Δηλαδή δεν λέει 2021 με 2026 ας πούμε. Δηλαδή μιλάμε για έναν ορίζοντα χωρίς ε, τέλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δείχνει και κάπως πώς πάντα πράγματα. Ο κύριος Άλλη μετά θα μας το πει, αλλά πιστεύω πως αυτή η κατάσταση δεν είναι σαφής και θα πρέπει αυτό να το θέσουμε επιτάπητος, ώστε να μην κάνουμε το λάθος, να υποχρηματοδοτήσουμε τις νέες μας φιλοδοξίες και μετά έχουμε και άλλες φιλοδοξίες. Άμυνα, μετανάστευση και τα προηγούμενα που είχαμε. Συνοχή που δίνει καλά αποτελέσματα. Η γεωργική πολιτική, την οποία προσπαθούμε να αλλάξουμε, ε, και να υποχρεώσουμε να αλλάξει η κοινή πολιτική γιατί έχει χάσει λίγο την ε, ορμή της. Αυτό που μας ανησυχεί λοιπόν, που έλεγε και ο κύριος Σαβάρμα, είναι η άμυνα δε είναι ένα θέμα το οποίο ε, μπορεί να ενταχθεί στο ΕΦΣΙ, στο ΕΦΣΙ 1 και στο 2 ε, και η δυνατότητα που έχουμε να δούμε, ε, να ελέγξουμε τα όσα μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα θα είναι όλο ένα και μικρότερη με τα blending και τις διάφορους τρόπους εγγυήσεις και τα λοιπά. Θα πρέπει λοιπόν ή να το ελέγξουμε ή αλλιώς να το ξεχάσουμε. Τώρα, αναπτυξιακή βοήθεια. Το, το σχέδιο για την Αφρική, συμφωνία με την Τουρκία, με τον ΟΗΕ, κάθε φορά να διακόπτει η πρόεδρος. Κοιτάξτε, δύο λεπτά είχα δώσει, δεν είχα δώσει επάπειρον. Κυρία Πρόεδρε, ε, αν δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε, σε λίγο θα είστε μόνοι σας εδώ. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δίνω το λόγο. Στον κύριο Φάρμπερ. thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σμιτ Φάρμπερ, ναι. Ναι, το όνομά μου είναι Σμιτ Φάρμπερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίαση των στοιχείων της εκθέσεώς του. Αποτυπώνει και τη δική μας λογική. Το σκεπτικό μας σε αυτό το έγγραφο εργασίας για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινήσαμε κι εμείς με το πλαίσιο του Brexit διότι είναι μια βασική πρόκληση την οποία θα αντιμετωπίσουμε στο επόμενο PDP, πώς θα καλύψουμε το κενό, εν μέρη με ίδιους πόρους, εν μέρη με νέες προτεραιότητες και, γι' αυτό και αναβάλαμε την πρότασή μας, θέλουμε επίσης να ξέρουμε τι ακριβώς θα συνεισφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τις παρελθούσες υποχρεώσεις τους και αυτό θα είναι σημαντικός παράγων για το μέγεθος του επομένου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στο έγγραφο που παρουσιάζει το σκεπτικό μας θα δείτε ότι μία βασική αρχή είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα είδατε ότι έχουμε βάλει ότι αν μια πολιτική δεν έχει προστιθέμενη αξία δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αν έχει μέση προς υψηλή θα πρέπει να ε, έχει κάποια συγχρηματοδότηση και αν έχει πάρα πολύ υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα έχει πλήρη χρηματοδότηση από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή πρέπει να είναι η κατευθυντήρια γραμμή για το επόμενο PDP και κάνουμε μια εσωτερική αναθεώρηση δαπανών για όλα τα προγράμματα. Εξετάζουμε βεβαίως και τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου Και όλα αυτά θα οδηγήσουν στις προτάσεις ανατομέα και στη συνολική πρόταση για το επόμενο PDP. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι η μεγαλύτερη χρήση οικονομικών εργαλείων και οικονομικών εγγύσεων. Πρέπει στο επόμενο PDP να είμαστε πιο ευέλικτοι θα πρέπει να αποφύγουμε το να κατανέμουμε εκ των προτέρων κάποια κονδύλια σε τόσο μεγάλο βαθμό στα κράτη-μέλη. Ίσως χρειαζόμαστε κάποια αποθεματικά προγραμμάτων που δεν θα έχουν κατανεμηθεί για να μπορούμε να αντιδράσουμε σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Και όσον αφορά τη διάρκεια, μπορούμε να έχουμε 5 ή 7 χρόνια ή πέντε συν με μια σημαντική αναθεώρηση στο ενδιάμεσο, ούτω ώστε να ευθυγραμμίζεται το PDP με την ε, γενικότερη κατάσταση. Ευχαριστώ. Για την γεωργική πολιτική, ποιο είναι το πρόγραμμά σας, γιατί μόλις ακούσαμε ότι εδώ παραμένει ένα παλαιό πρόγραμμα. Έχετε σκεφτεί κάτι όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας. Ο κύριος Σμιτ Φάρμπερ. Κοιτάξτε, τώρα μόλις ξεκινάμε να ασχολούμεθα με τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ λύσεις ε, για μεταρρυθμίσεις και στις γεωργικές πολιτικές. Δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένα για προγράμματα ε, συνταξιοδότησης. Αλλά ε, όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε. Ο κύριος Τάραντ είχε ζητήσει το λόγο και η κυρία Γιάλα Σέντερ. Θα είμαι πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σάρπαμα που μας παρουσίασε αυτή την έκθεση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και τον Αύγουστο θα σας στείλω ένα email με τις τέσσερις αρχές και θα τονίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και επισκοπήσεις και αξιολογήσεις και όλα αυτά τα οποία θα έχουν βασική και σε επιπτώσει στο έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυρία Γιάλα Ζέντερ. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, κάτι σχετικά με την ε, πρόταση για την άμυνα. Γιατί η ιδέα που είχαμε όταν είπαμε ότι η άμυνα μπορούσε να αποτελέσει προστιθέμενη αξία ήταν ότι θα γινόταν οικονομίες κλίμακας. Ότι δηλαδή τα όσα δαπονώνται σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να δαπονηθούν σε ευρωπαϊκό και να μπορέσουμε να ζητήσουμε να από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που κάθε ε, ε προπολογισμό, ο οποίος κάθε φορά γίνεται και πιο ισχνός, να βάλει και κάτι παραπάνω για να χρηματοδοτηθεί αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη ένα κομμάτι από αυτά που δαπανούν κάθε χρόνο ο καθένας στο δικό του προπολογισμό να τα βάλουν σε ένα κοινό ε, κορβανά ώστε να αρχίσει με αυτόν τον τρόπο η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. δεν δίδονται χρήματα χωρίς ε, αρμοδιότητες. Μπορούμε να ε, ε, χρηματοδοτήσουμε το μίσο που έχουμε αρμοδιότητα. Πώς να χρηματοδοτήσουμε πολιτική άμυνα αν δεν έχουμε σχετικές αρμοδιότητες. Θέλετε το λόγο. Ο κύριος Σμιτ Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, συμφωνώ. Πρέπει να δούμε τι μας επιτρέπει η συνθήκη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Παρόλα αυτά, στα θέματα της έρευνας για την άμυνα ή της ανάπτυξης πρωτοτύπων, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Και αυτό θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα για τα κράτη-μέλη αν γίνονται αυτά συνολικά από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό να γίνει μια κοινή ανάπτυξη πρωτοτύπου από τα κράτη-μέλη, εξοικονομώντας χρήματα από τους μεμονωμένους προϋπολογισμούς. Βεβαίως, λέει η Πρόεδρος. θα πρέπει να επιλέγονται τα έργα με βάση ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχε αρμοδιότητε. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό χωρί να υπάρχει αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο τομέα. Συνάδελφο Σαρβάμα. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προσπαθήσω να απαντήσω προς τους ε, σκιώδεις συζητητές, ε, προς τον κύριο Άλλη ε, που ανέφερε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα εκφώνησης προϋπολογισμού. Όντως, και εγώ το έχω συζητήσει αυτό το θέμα, θα πρέπει να έχουμε ένα κύκλο στον προϋπολογισμό. Ο κύριος Λιμπεράτσκι δεν είναι πια μαζί μας. Συμφωνώ όμως απολύτως με αυτά που είπε. για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα που θα πρέπει να συμβαδίζει με την ιεράρχηση των ε, μέτρων και για την πολιτική συνοχή και κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να δούμε πώς θα το οργανώσουμε καλύτερα και τα δύο. Για τη συνοχή έχω κάποια σχέδια Θα δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η δομή των δαπανών. όταν θεωρούμε ότι επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα επιτυχή αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. κατά πόσο μπορούμε με τον εξυγχρονισμό να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αντί να συνεχίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Ευχαριστώ και την κυρία Γιάλα Σέντα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβασή σας. Αν σωστά σας κατάλαβα, συμφωνώ πολύ τους μαζί σας, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε με μία προϋπάρχουσα ιδέα ότι πρέπει να δεχθούμε ένα χαμηλό προϋπολογισμό, να μην υποκύψουμε λοιπόν σε αυτή την προκατάληψη. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις με τα σύνορα, με τη μετανάστευση, με την άμυνα. Και παράλληλα τα κράτη-μέλη αυτό που λένε από τη μία, από την άλλη το παίρνουν πίσω. Θα πρέπει τα χρήματα που διαθέτουμε το προϋπολογισμό, τα διαθέτουμε για αυτό το οποίο λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε. Θα είχα πολλά να σας πω, αλλά δεν έχω το χρόνο. Αν έχετε την καλοσύνη, στείλτε μου email με τις προτάσεις σας. Όπως μου υποσχέθηκε ήδη ο κύριος Τάραντ, θα μου το στείλει τον Αύγουστο. Μέρα παραμέρα θα περιμένω να μου στέλνετε email στις διακοπές μου. Και στις 13 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιούγκερ, θα μας κάνει ίσως την πιο σημαντική ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης και ίσως εκεί προκύψουν κάποιες ιδέες να δούμε αν συμβαδίζουμε με τη γραμμή που θα έχει χαράξει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, το 14, μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Ο κύριος Άλλη θα μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα ε, των πόρων είναι πολύ σημαντικό. Είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την Ένωση. Παρότι είναι γενικώ ανεπαρκής, η παρακολούθηση της δαπάνης των ιδίων πόρων ε, και αν και κατά πόσον δαπανώνται σημαντικά και ε, ουσιαστικά και αποτελεσματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχουν και τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες ε, ο προϋπολογισμός στηρίζει τις κοινέ πολιτικές και τους στόχους και προσφέρει κεφάλαια κίνησης για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Βασικός στόχος ε, του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να είναι υποστήριξη ταχύτερη μεγέθυνση στις λιγότερο ανεπτυγμένε περιφέρειες για να επιτευχθεί ισοδύναμο επίπεδο ανάπτυξης σε όλα τα κράτη-μέλη και ως εκ τούτου θα πρέπει να μπορούμε να υποβάλουμε ε, αρκετές προτάσεις στις αρμόδιες επιτροπές. Καταρχήν, ε, η κατανομή των πόρων επικεντρώνεται σε τομείς όπου είναι απαραίτητη η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ότι μπορεί να δημιουργηθεί υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Παραδείγματο χάρη η έρευνα και ανάπτυξη, όπως επίσης και ε, ε, θέματα που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Δεύτερον, μακροπρόθεσμη ωφέλη θα πρέπει να δαπανώνται σε τομείς που είναι μακροπρόθεσμα υποφελείς και όχι αυτούς που ε, βραχυπρόθεσμα μόνο έχουν ωφέλη. Ως εκ τούτου θα πρέπει ένα μέρος του προϋπολογισμού να ε, δαπανάται σε θέματα που φορούν την κλιματική αλλαγή. Ε, μακροπρόθεσμη στόχοι. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει σημαντικό ρόλο στο στόχο των διαδοχικών πολιτών ε, δημοσιονομικών πλαισίων για το 2020 ο ορίζοντας του 2020 πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως επίσης και οι 10 προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker. Ε, ε, πιστεύουμε επίση ότι απλούστεροι και σαφέστεροι κανόνες θα συμβάλλουν στην ταχεία κατανομή των πόρων και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Ενώ ταυτόχρονα ο τρόπος ε, μέτρηση της κατανομής των κονδυλίων θα πρέπει να βελτιωθεί και να δώσει έμφαση σε έργα που, τα οποία θα είναι εποφελία όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παρέχουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. danke, Frau Ευχαριστούμε κυρία Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Αλή για την ε, πρότασή του. σχετικά με το σύστημα ιδιών πόρων. Υπάρχει ένα σημείο ε, που δεν μου ήταν σαφές, το σημείο 10 λέει ε, πολιτικές που θα ωφελήσουν όλους τους πολίτες. Λέει ποια πρέπει να είναι η μέθοδος μέτρησης της αξίας των έργων. και θα ήθελα να δω πώς λαμβάνουμε υπόψη και τις πιο μακροπρόθεσμες πολιτικές. Έχουμε συνηθίσει τις βραχυπρόθεσμες πολιτικές, αλλά οι μακροπρόθεσμες νομίζω καλύπτουν τη γεωργία και τη συνοχή. Uh, concentrating on the revenue side of the budget. Uh, of course, thinking Μιλάμε για τον καλύτερο τρόπο της χρήσης των δαπανών και σκεφτόμαστε τον πόρων και σκεφτόμαστε τις δαπάνες. Όμως, με βάση το σύστημα εισόδων που υπάρχει, πρέπει να παραδεχτούμε ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και πολύ σοβαρό. Το παρόν σύστημα εσόδων παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες. Στο έγγραφο που αφορά το μέλλον της ε, χρηματοδότησης της Ένωσης που, παρήχει, που παρουσίασε η Επιτροπή ε, πριν από δύο εβδομάδες γίνεται αναφορά στην έκθεση του, του Δεκεμβρίου 2016 της, της ε, ε, υψηλής ε, ομάδας για την παρακολούθηση των εσόδων και αναφέρεται ότι το τωρινό σύστημα είναι εξαιρετικά αδιαφανές, σύνθετο και γεμάτο δυσκολίες. Είναι πολύ σύνθετο. Υπάρχουν το 70% των εισφορών των κρατών μελών ε, έναντι των πραγματικών ιδίων πόρων. Ως εκ τούτου, η απόφαση του 1970 για την εισαγωγή ενός συστήματος ιδίων πόρων για να ενισχυθεί η ε, οικονομική ανεξαρτησία της τότε κοινότητας υπονομεύεται σοβαρά. Το πρόβλημα συνίσταται πολύ ενοχλητική θα έλεγα κατάσταση που δημιουργείται με, με το τρέχον σύστημα όπου έχουμε εισφέροντες και ε, ε, ε, δικαιούχους κατά κάποιο τρόπο οι οποίοι τελικά ανταγωνίζονται μεταξύ τους με μηδενικό αποτέλεσμα πολύ συχνά. Υπάρχει αυτή η γενική αντίληψη ότι πρέπει να υπάρχει το λεγόμενο juste retour, δηλαδή η σωστή δίκαιη επιστροφή που αυτή τη στιγμή είναι ένας αριθμητικά απλός τρόπος για την αντιστάθμιση των δαπανών στον τομέα ε, με τις εθνικές ε, εισφορές. Το σύστημα τώρα δείχνει ότι αυτή όχι απλουστευμένη αλλά απλουστευτική ε, προσέγγιση με την οποία τα κράτη-μέλη ε, αντιμετωπίζουν την συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό είναι στριβλή. Διότι πολλές πλευρές της σχέσης μεταξύ εθνικού και κοινοτικού προϋπολογισμού μπορούν να ειδωθούν με αυτόν τον ε, απλουστευτικό τρόπο. Επίσης υπάρχει το, θέμα, το σύστημα των επιστροφών που ξεκίνησε με τις επιστροφές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά έχουμε επιστροφές επί επιστροφών που μεγαλώνουν. Αυτές έχουν αποτελέσει αντικείμενο μη διαφανούς συζήτησης αν αισθάνεστε ότι μακρηγορώ, θα σταματήσω στο σημείο αυτό, λέει ο μιλητή. Είπαμε δύο λεπτά ε, καταρχήν. Δεν το γνώριζα, δεν το γνώριζα. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εκπροσωπώ τον σκιώδιο εισηγητή μας, τον κύριο Τεκόφσκι. Μου έχει δώσει υλικό που θα ε, χρειαστεί πέντε λεπτά για να το διαβάσω. Έτσι λοιπόν θα αναφερθώ μόνο στα βασικά σημεία. Ο σκιώδης, ο κύριος Τεκόφσκι, συμφωνεί με τον κύριο Πυρίνσκι ότι το τρέχον σύστημα είναι εντελώς ξεπερασμένο, υπερβολικά σύνθετο και ε, του λείπει διαφάνεια. Ως εκ τούτου, μια σε βάθος μεταρρύθμιση είναι όντως απαραίτητη το θέμα είναι με ποιο τρόπο, βεβαίω πώς θα γίνει η αλλαγή αυτή. Και οι προτεραιότητες είναι η επάρκεια, διαφάνεια, σταθερότητα, απλότητα, ξεκάθαρη, ε, ξεκάθαρη εικόνα, χαμηλό κόστος λειτουργίας, ευρωπαϊκή ε, προστιθέμενη αξία και ένα σύστημα που θα είναι κατανοητό από τους Ευρωπαίους ε, φορολογούμενους. Ο Σκιώδης Ομιλητής τη συμφωνεί με τις προτάσεις της ομάδας ψηλού επίπεδου για τις ιδίους πόρους, για τη διατήρηση των παραδοσιακών ιδίων πόρων, αλλά να, για, υπέρ της απαλλαγής από τον διορθωτικό μηχανισμό που στηρίζει, το, τρέχον σύστημα ιδίων πόρων θα πρέπει να αντικατασταθεί με το σωστή μεταφορά του σωστού επίπεδου του ΦΠΑ από τις, τα κράτη-μέλη και άλλους πόρους που θα προέρχονται από ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν νέοι ήδη πόροι. Όλο αυτό, όλο, όλοι το έχουμε αυτό κατά ο σκιώδης ομιλητής, οι σκιώδεις ομιλητές και εγώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο, Όλη για, τον κύριο Αλή για το έργο του. Ο σκιώδης ομιλητής ε, ε, αναφέρει ή προτείνει μάλλον να γίνει μια συνάντηση σκιωδών ε, εισηγητών ώστε να επιληθεί το θέμα της γνωμοδότησής σας όπου αναφέρεται, που, όπου κατά τη γνώμη του θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα, ένα ξεκάθαρο θέμα για τα έσοδα. Το κομμάτι αυτό δηλαδή της γνωμοδότησης πρέπει να ενισχυθεί κατά τη γνώμη τους. Επίσης το θέμα των δαπανών και της κατανομής τους αυτό το, το αναφέρεται. Το θέμα όμως των εσόδων τους απασχολεί. Αυτά είχα να πω νομίζω. Ευχαριστώ. Dankeschön. Wir sind da im Moment noch nicht richtig auf Ballhöhe, ne? das muss ich schon mal sagen. Da sind wir auch noch nicht konkret genug. Ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο Τάρανα το λόγο, δύο λεπτά, όχι περισσότερα. One. Uh, I, uh, agree. Συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια και τις ερωτήσεις, αλλά κύριε Άλλη, μην πυροβολείτε τον ε, αγγελιοφόρο. Έχω να πω κάτι εκ μέρους του Σκιώδους, που λέει ότι είναι μια πράσινη δήλωση ε, αυτή εδώ και βρίσκω ότι αυτή η ε, έκθεση είναι ακατάλληλη. Θα έπρεπε να την αναβάλουμε και να συντάξουμε μία πλήρως νέα έκθεση. Εάν δεν το επιτύχουμε αυτό, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε άλλα βήματα. Αυτά λοιπόν λέει ο δικός μας κοιόδης ηγητής προς ενημέρωσή σας. Um ναι, δεν είναι πολλά τα στοιχεία σχετικά με τους ιδίους πόρους αυτή η γνωμοδότηση, όντως θα βρουν οι με τον εισηγητή μία λύση για να μην υπάρξει όξυνση του θέματος από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Μοντάνια. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Να σχολιάσω κάποια από τα θέματα που αναφέρονται στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, και να αντιδράσω και σε κάποια από τα σχόλια των συναδέλφων για την προστιθέμενη αξία καταρχήν. Όντως, ε, τονίζεται και στην προηγούμενη έκθεση που ακούσαμε για το PDP. Και αναφέρθηκε και στο έγγραφο της Επιτροπής που αναφέρθηκε προηγουμένως. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σαφώς και πρέπει να είναι το στοιχείο που μας καθοδηγεί για να καθορίσουμε το ποια προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα και ε, προσθέμενη αξία μπορεί να βρεθεί και από την πλευρά των εσόδων σύμφωνα με την έκθεση Μόντι και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο εξετάζουμε. Δεν ε, ε, ήταν ένα στοιχείο που λαμβάναμε υπόψη στο παρελθόν. Δηλαδή, το σκεπτικό είναι γιατί να μην χρησιμοποιούμε τους ίδιους πόρους, νέους ίδιους πόρους, για να έχουμε σύνθετα κέρδη και να υποστηρίξουμε κάποιους από τους στόχους της πολιτικής μας. Μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ε, η μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Ε, υπάρχουν ε, λοιπόν δυνατότητες οι ίδιοι να χρηματοδοτούν αυτούς τους στόχους και όχι μόνο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο σημείο που τονίσατε είναι η μεθοδολογία της καθαρής ισορροπίας να εξηγήσουμε γιατί αυτό αποτελεί πρόβλημα και στην έκθεση Μόντι και στο έγγραφο με το έγγραφο προβληματισμό της Επιτροπής αναφέρεται ότι με το net balance έχουμε κυρίως ε, τα θέματα δαπανών, ιδίως στη γεωργία και στη συνοχή. Οι δαπάνες που έχουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία δεν αναγνωρίζονται με αυτή τη μέθοδο και αυτό έχει ε, ως συνέπεια το ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, το υποστηρίζουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια μεγάλη επιχορήγηση για έρευνα θα υπολογιστεί με τη μεθοδολογία αυτή ως κάτι το οποίο υποφελείται ε, επωφελείται το, το Πανεπιστήμιο που είναι ο κύριος φορέας για αυτή την επιδότηση. Θεωρείται ο δικαιούχος στο Λουξεμβούργο, εν, σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ενώ επωφελούνταν πέντε ή έξι πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη από την ίδια επιδότηση για την έρευνα. Το ίδιο και για την εξωτερική ασφάλεια. Πολλά από τα χρήματα που δίδονται για την προστασία των εξωτερικών συνόρων θεωρούνται κέρδος για την Ελλάδα και κόστος για όλες τις άλλες χώρες. Γι' αυτό η μέθοδος δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική και προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα της μεθοδολογίας του καθαρού υπολείπου. Άλλο ένα σχόλιο για κάτι που δεν αναφέρεται στη γνωμοδότηση, αλλά αναφέρθηκε σε σχέση με τις επιστροφές. Μπορεί στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής να το έχετε δει. Είναι ξεκάθαρη η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει ε, να απαλλαγούμε από το σύστημα αυτό και να βρούμε ένα σύστημα πιο διαφανές και απλούστερο. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσαμε. Νομίζω ότι τον προϋπολογισμό δεν μπορούμε να τον βλέπουμε μόνο ως δαπάνες. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Όσο για την πολιτική συνοχής, πρέπει να την δούμε μακροπρόθεσμα και ευχαριστώ να οργανώσω μια συνάντηση με τους σκιώδεις συζητητές ε, πριν από την ε, εκπνοή των προθεσμιών βεβαίως και θα έλεγα να βάλουμε ως προθεσμία την 30 Οκτωβρίου και στην Επιτροπή μας να γίνει ψηφοφορία στις 22 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η πρότασή μου. Θα ήθελα να μου στείλετε email με τις προτάσεις και είμαι ανοιχτός για τις προτάσεις που θα λάβω. Σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο σημείο 15, υλοποίηση των διαφορετικών ταμείων 2007-2013. Έργα προτεραιότητας στην Ελλάδα. τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Υπάρχουν 81 έργα προτεραιότητα. Το 2015 το Σεπτέμβριο επισκεφθήκαμε ε, νομίζω 7 από αυτά στην Ελλάδα και θα θέλαμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει με όλα τα υπόλοιπα ε, έργα, ποια είναι η κατάσταση, τι έχει ολοκληρωθεί, τι χρηματοδοτείται, τι δεν πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται και γι' αυτό έχουμε καλέσει εδώ το Γενικό Διευθυντή Μαχλεμέτ, δεν τον βλέπω όμως ακόμη. Εμείς τον είχαμε προσκαλέσει. Σας υπενθυμίζω ότι χρηματοδοτούμε 100% τα έργα αυτά κατά την περίοδο αυτή και έχουμε σαφώς λόγους να ασχοληθούμε με τον έλεγχο του προϋπολογισμού και γι' αυτό το βάλαμε στην ημερήσια διάταξη και γι' αυτό θέλαμε να έχουμε... Α, καλώς ήρθατε κυρία Γενική Διευθυντά. Ich habe die Kollegen schon äh, über die bisher, bisherigen Geschehnisse Ενημέρωνα λίγο του συναδέλφου για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, κύριε Λεμέτ. Χαιρόμαστε που ήρθατε στην Επιτροπή μα και σα δίνουμε αμέσω το λόγο για να μα πείτε τι έχει γίνει με τα 181 έργα προτεραιότητα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Εμεί είχαμε επισκεφθεί 7 από τα έργα αυτά και θέλουμε ε, να έχουμε μια συνολική εικόνα της προγραμματικής περίοδου για την Ελλάδα διότι πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων, αφού μιλάμε για χρηματοδότηση 100%. Έχετε το λόγο, κύριε Γενική Διευθυντά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι και κύριοι βουλευτές, καλή σας μέρα. Χαίρομαι που είμαι σήμερα στην Επιτροπή σας, διότι θα ήθελα να σας ενημερώσω κυρίως για δύο πολύ σημαντικά συνεχιζόμενα προγράμματα δράσης. Θα τα γνωρίζετε οπωσδήποτε. Το πρόβλημα με τα σχέδια δράσης είναι ότι υιοθετούνται και μετά ξεχνιούνται. Εδώ όμως είναι, πιστεύω, αρκετά σημαντικά τα θέματα, ούτως ώστε να τα παρακολουθούμε τακτικά με την απαιτούμενη φροντίδα. Τα δύο σχέδια δράσης αφορούν δύο τομείς που αποτελούσαν παραδοσιακά την αχίλιο πτέρνα της πολιτικής συνοχής όσον αφορά ε, τα ποσοστά σφάλματος, τις κρατικές συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. Και στους δύο αυτούς τομείς, το ποσοστό σφάλματος σαφώς είχε σχέση με ελλείμματα διοικητικής ικανότητας σε διάφορα επίπεδα στα κράτη-μέλη. και αυτό αφορούσε τις δομές ε, που υλοποιούσαν τα έργα της πολιτικής συνοχής και πιο πρόσφατα τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Τα σχέδια δράσης επικεντρώνονται σε αυτή την πτυχή του προβλήματος, στο πώς να βοηθήσουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν διοικητική ικανότητα σε αυτούς τους τομείς, ούτω ώστε τα ποσοστά ασφάλιματος να είναι πολύ μικρότερα από ό,τι στο παρελθόν. Ένα πρώτο πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα προέκυψε από τα ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου για το 2015. Οι πρώτες τρεις πηγές φάλματος στην πολιτική συνοχής σταμάτησαν να παρουσιάζουν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και οι δημόσιες συμβάσεις και οι κρατικές ενισχύσεις δεν ήταν πλέον μέσα στα τρία πρώτα όσον αφορά τα ποσοστά σφάλματος. Τα ευρήματα λοιπόν του ελεγκτικού συνεδρίου μας έδειξαν ότι η συχνότητα σφάλματος και στους δύο αυτούς τομείς είχαν μειωθεί σημαντικά και χωρίς ε, να ξέρουμε τα αποτελέσματα για το 2016 ε, πιστεύουμε έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι δεν ε, ήταν ένα φαινόμενο που μόνο μια χρονιά εμφανίστηκε το 2015 αλλά πιστεύουμε ότι αυτή η σημαντική βελτίωση θα επιβεβαιωθεί και για το 2016. Αυτό ελπίζουμε. Έχω ετοιμάσει και κάποιες διαφάνειες, τις οποίες αρχίζω να σας παρουσιάζω, ξεκινώντας με τις ε, δημόσιες συμβάσεις και το σχέδιο δράσης σχετικά με αυτό. Για αυτό το σχέδιο δράσης, όπως και για τις κρατικές ενισχύσεις, πολύ μεγάλη σημασία έχει ο νέος μηχανισμός που έχουμε για την περίοδο 2014-2020, την ε, εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις σε ορισμένους τομείς από τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις πληρωμές στα εν λόγω κράτη-μέλη και για τους εν λόγω τομείς. Την άνοιξη του 2017 κάναμε ήδη μια προκαταρκτική εξέταση των αποτελεσμάτων αυτού του μηχανισμού αιρεσιμότητας που έδειξε πολύ θετικά στοιχεία ιδίως για τις κρατικές συμβάσεις και για τις κρατικές ενισχύσεις. Πιστεύω ότι η εκ των προτέρων ερεσιμότητα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που οθεί τα κράτη-μέλη να εστιάσουν στη βελτίωση της ικανότητάς τους σε αυτούς τους τομείς. Για την περίοδο 2014-2020, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε τέσσερις δημόσιες συμβάσεις και 12 ε, κράτη-μέλη που έπρεπε να βελτιώσουν στοιχεία με βάση την αιρεσιμότητα. Τώρα, τέσσερα κράτη-μέλη ε, παραμένουν, δηλαδή τα οκτώ κράτη-μέλη βελτίωσαν την κατάσταση. Και ακόμη και για τα τέσσερα κράτη-μέλη που απομένουν, οι προοπτικές φαίνονται καλές και ελπίζουμε ότι για τα περισσότερα, αν όχι για όλα, δεν θα χρειαστεί να αναστείλουμε πληρωμές, διότι θα έχουν κάνει αυτά τα οποία τους έχει ζητηθεί να κάνουν. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο σε αυτό το σχέδιο δράσης είναι η ομάδα εργασίας για τις κρατικές συμβάσεις. Μια ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε το 2014 στην Επιτροπή συμπεριλαμβάνει όλους τους ενδιαφερομένους, τη Γενική Διεύθυνση για τα επενδυτικά και Διαφθορτικά ταμεία, όπως και η Γενική Διεύθυνση Grow και με υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτή η ομάδα εργασίας έχει τρεις τομείς δράσης. Πρώτον, να τηρούνται οι κοινοτικές οδηγίες για τις ε, κρατικές συμβάσεις, μια συνεχιζόμενη πρόκληση και θα επανέλθω σε αυτό, διότι υπάρχει και μια νέα οδηγία τώρα για τις κρατικές συμβάσεις, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ και θεωρητικά θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη μέχρι τα μέσα του προηγουμένου έτους, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αυτή η διαδικασία. Δεύτερο τομέα δράση αυτή τη ομάδα εργασία είναι η ενίσχυση τη αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στι διαδικασίε κρατικών συμβάσεων. Μια νέα διάσταση που δίνεται από αυτή τη νέα οδηγία που ανέφερα. Ενθαρρύνουμε τη χρήση των κρατικών συμβάσεων ως εργαλείο στρατηγικής. Δηλαδή να μην ζητείται μόνο ο, ο μειοδότης, αλλά στην προκήρυξη του έργου να συμπεριλαμβάνονται κάποια στοιχεία περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα ή καινοτομίας και τα αναφέρω αυτά εν είδη παραδείγματος. θέλουμε να εφαρμοστούν όλα αυτά όσο το δυνατόν ευρύτερα στην πολιτική συνοχή στο μέλλον, ούτω ώστε οι κρατικές συμβάσεις να μην λαμβάνουν υπόψη μόνο το χαμηλότερο κόστος, αλλά να έχουν μια συνεκτική, ολοκληρωμένη εικόνα ε, των αποδοτικών έργων. Κάτι που θέλω να αναφέρω ως ε, αποτέλεσμα αυτής της ομάδας εργασίας είναι ένας οδηγός που έτυχε εξαιρετική αποδοχή στα κράτη-μέλη και τον χρησιμοποιούν στα κράτη-μέλη. Το βλέπουμε από τον αριθμό ε, οδηγών που έχουν ε, κατεβάσει από το διαδίκτυο τα κράτη-μέλη. Ένας εκτενέστατος οδηγός με πολύπλοκους κανόνες που όμως είναι και απλές οι οδηγίες του για να αποφεύγονται οι συνηθισμένες ε, οι συνηθισμένες παγίδες τις οποίες πέφτουν αυτοί που εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα. Θέλουμε να επικαιροποιήσουμε αυτόν τον οδηγό και ελπίζουμε ότι πριν τα τέλη του έτους θα έχουμε την επικαιροποιημένη εκδοχή του οδηγού αυτού στο διαδίκτυο. Θέλω επίσης ε, να σας αναφέρω τι έχουμε κάνει για συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Έχουμε ακολουθήσει μια πολύ πρακτική προσέγγιση και είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την πολύ πρακτική προσέγγιση. Χρησιμοποιούμε τον προϋπολογισμό μας για τεχνική βοήθεια και ε, έχουμε ζητήσει και από ένα τρίτο φορέα, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον ΟΣΑ, να βοηθήσει συγκεκριμένα τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία ούτως ώστε να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στη Σλοβακία με τη δημιουργία μιας στρατηγικής ηλεκτρονικών συμβάσεων. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα αυτής ε, της ε, συγκεκριμένης λύσης που βρέθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένες χώρες σε αυτό το slide, σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τη συνεργασία μας με τον ΟΣΑ για την Βουλγαρία και τη Σλοβακία. Μια άλλη πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο αφορά το Σύμφωνο Ακαιρεότητας. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και το υλοποιούμε με την τεχνική μας βοήθεια. Έχουμε ως εταίρο τη Διεθνή Διαφάνεια, μια μη κυβερνητική οργάνωση, και επιβλέπει εθελοντικά διάφορες διαδικασίες κρατικών συμβάσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι διότι αρκετά κράτη-μέλη έχουν επωφεληθεί αυτή της ευκαιρίας. Βλέπετε στη διαφάνεια 11 κράτη-μέλη που έχουν ζητήσει τη βοήθεια της διεθνούς διαφάνειας. Είναι ένα πιλωτικό έργο το οποίο καλύπτει 17 έργα στα 11 κράτη-μέλη. Και αυτό που θα θέλαμε είναι όλοι οι συμβαλόμενοι στη διαδικασία κρατικών ε, συμβάσεων ε, να προσυπογράψουν ένα κώδικα δεοντολογίας, ούτως ώστε να υπάρχει ένας εξωτερικός επόπτης, η διεθνής διαφάνεια, που θα διασφαλίζει ότι τηρούνται οι απαιτούμενοι όροι από όλους τους συμβαλωμένους, από τον οργανισμό που κάνει την προκήρυξη και από αυτούς που υποβάλλουν προσφορές. Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω αφορά πιο συγκεκριμένα την απάτη. Ευτυχώς είναι οριακό φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εντοπίζουν συγκεκριμένες ε, υποθέσεις απάτης και να τις καταπολεμούν καλύτερα. Έχουμε ένα εργαλείο πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα ε, εργαλείο εξόριξης δεδομένων, που προσπαθεί να εντοπίσει ύποπτα στοιχεία σε κάποια διαδικασία κρατικών συμβάσεων. Ένα εργαλείο που αναπτύξαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διαθέτουμε δωρεάν στα κράτη-μέλη και πάλι βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη το ε, έχουν ζητήσει, πολλά κράτη-μέλη μας έχουν ζητήσει να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο πληροφορικής Ενθαρρυντικό λοιπόν αυτό, διότι βοηθά τα κράτη-μέλη να εντοπίσουν κάποιες ε, ύποπτες ε, συνθήκες σε μια διαδικασία κρατικών προμηθειών, κρατικών συμβάσεων, για να μπορέσουν ε, να στοχεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου καλύτερα. Θέλω τέλος ε, να σας παρουσιάσω και μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης, την οποία συνεχίζουμε και για τις υποψήφιες χώρες. Είναι η πρωτοβουλία ΤΑΙΕΚΣ και η αρχή του ΤΑΙΕΚΣ είναι ότι βρίσκουμε εμπειρογνώμονες μέσα στα κράτη-μέλη, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τις διοικήσεις άλλων κρατών μελών να βελτιώσουν την τεχνογνωσία τους. Λειτουργεί πολύ καλά αυτό το σύστημα. Έχουμε αρκετές ανταλλαγές και πολλές δράσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής και σε μεγάλο βαθμό Έχουμε εμπειρογνώμονε σε θέματα κρατικών συμβάσεων που βοηθούν επιτόπου άλλα κράτη-μέλη, άλλα υποψήφια κράτη-μέλη. Συμμετέχουν 21 ε, κράτη. Δεν επαναπαυόμαστε όμως. Ελπίζουμε ότι θα επιβεβαιωθεί η θετική τάση όσον αφορά τη βελτίωση στις κρατικές συμβάσεις. Αλλά ξέρουμε ότι είναι και λίγο έργο σύσυφου αυτό το οποίο κάνουμε. Υπάρχει νέα οδηγία που δεν έχει ακόμη περάσει σε εθνικό δίκαιο σε όλα τα κράτη-μέλη. Παραμένουμε λοιπόν σε επαγρύπνηση. Παρακολουθούμε το θέμα και όπως σας είπα τον οδηγό που έχουμε βάλει στο διαδίκτυο θα τον επικαιροποιήσουμε για αυτούς που ασχολούνται με τις κρατικές συμβάσεις. Να σας πω ακόμη ότι με τη νέα οδηγία υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούνται οι κρατικές συμβάσεις με πιο στρατηγικό τρόπο. Αυτό επιδιώκουμε. Και όσον αφορά το σχέδιο δράσης, βεβαίως και θα παρακολουθούμε την σωστή υλοποίησή του μαζί με τη Γενική Διεύθυνση GROW και τους αρμόδιους επιτρόπους, τις επιτρόπους ε, Κρέτσου και Βιενκόφσκα. Τώρα περνώ στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Οι προκλήσεις είναι οι ίδιες. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη διοικητική ικανότητα και μας ενδιαφέρει διπλά το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, διότι όχι μόνο φύγεται ο κρατικός προϋπολογισμός, μπορεί να χορηγούνται περισσότερο, περισσότερες κρατικές ενισχύσεις από ό,τι θα επέτρεπαν οι κανονισμοί. Αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνουμε και το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό είναι ότι λόγω του φόβου της πολυπλοκότητας των κρατικών ενισχύσεων πολλές εθνικές αρχές ε, προτιμούν να ακολουθούν τον κανόνα de minimis, δηλαδή προσπαθούν να βρίσκουν κάποιο τρόπο να ξεφεύγουν από τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων για να μην διατρέχουν κανένα κίνδυνο όσον αφορά ε, την πολυπλοκότητα του συστήματος. Αλλά αυτό δεν μας εγγυάται ότι η προσέγγιση που ακολουθούν είναι η καλύτερη. Ότι επιτυγχάνονται δηλαδή οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, να βελτιώσουμε και τα έγγραφα τα οποία εκδίδουμε, όπως αυτό που έκδοσαμε τον Ιούλιο του 2016 με διευκρινιστικά στοιχεία για την έννοια των κρατικών ενισχύσεων. Σίγουρα όμως μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα. Έχουμε θετικά στοιχεία για την αιρεσιμότητα. Εδώ λιγότερα κρατημέλη είχαν εξ αρχής κάποιες ελλείψεις. Ε, η Ιταλία είναι η μόνη από τις πέντε χώρες που αρχικά είχαν ελλείψεις και συνεχίζει να έχει κάποιες ελλείψεις και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρει τελικά. Έχουμε και θετικά παραδείγματα να σας αναφέρουμε. Να τονίσουμε καταρχήν πώς ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση ε, σε περιορισμούς Κάθε κράτος μέλος μπορεί να κάνει ένα μητρό για τον κανόνα de minimis, διότι η δυσκολία με τον de minimis είναι ότι μπορεί να περάσεις πάνω από το maximum που είναι 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια, αν ως εταιρεία πάρεις πέντε φορές από 50.000 ευρώ. Για να το καταγράψεις αυτό χρειάζεσαι μια κεντρική βάση δεδομένων για να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει μία εταιρεία που με πολλές de minimis ενισχύσεις ξεπερνάει το συνολικό κατόφλι. Το ελεγκτικό συνέδριο πρότεινε να εφαρμόσουμε σε κάθε κράτος μέλος ένα κεντρικό μητρό. Προτείναμε και σχετική νομοθεσία, αλλά ε, δεν έγινε αποδεκτό. Αυτό που κάναμε εμείς μέσω της ε, εκ των προτέρων ερεσιμότητας είναι από κάποια κράτη-μέλη να αποσπάσουμε τη δέσμευσή τους ότι θα δημιουργήσουν τέτοιο κεντρικό μητρό σε επίπεδο κράτους μέλους και αυτό έχει γίνει στην Τσεχία και στη Σλοβακία, πράγμα που μας ικανοποιεί ιδιαίτερος. συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο και Κοντ για να, να στοχεύουμε τους τομείς εκείνους όπου έχουμε περισσότερες κρατικές ενισχύσεις και όπου είναι και πιθανότερα τα σφάλματα. Στην έρευνα και καινοτομία, σε δράσεις ευρείας ζώνης, και σε ενεργειακά έργα. Και μαζί με την Γενική Διεύθυνση ΚΟΜΠ έχουμε οργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για πολλά κράτη-μέλη για τα συγκεκριμένα αυτά θέματα όπου υπάρχουν πολλές κρατικές ενισχύσεις. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο όμως και στις κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία όπως και στις κρατικές συμβάσεις. Πάλι έχουμε το σύστημα TAIEX ε, για ενημέρωση από εμπειρογνώμονες. Και ένα τελευταίο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω για τις κρατικές ενισχύσεις είναι ότι πιστεύουμε ότι έχουμε επιτύχει μια πραγματική επανάσταση στην Ελλάδα. όχι μόνο με την οικονομική ενίσχυση που παρέχουμε, αλλά και με την τεχνική βοήθεια. Και μαζί με την Υπηρεσία Στήριξης Διαφορετικών Μεταρρυθμίσεων, Έχουμε τώρα ένα σύστημα πληροφορικής στην Ελλάδα που δίνει ισχυρές εγγύησεις που ήταν απολύτως απαραίτητες για θέματα κρατικών ενισχύσεων. Ούτε ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανότητα διαφθοράς και απάτης. Κλείνοντας λοιπόν την παρουσίασή μου, Πρόεδρε, Θέλω να σας πω ότι ε, ενθαρρυνόμενοι από τα πρώτα θετικά αποτελέσματα συνεχίζουμε ακάθεκτοι Δεν επαναπαυόμαστε καθόλου, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση και με τα χαράς θα επανέλθουμε για να σας ε, περιγράψουμε την πρόοδο που ελπίζω ότι θα έχει επιτευχθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Και ελπίζω ότι θα το επιβεβαιώσουν και τα ετήσια ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Στην αρχή δεν είμαι σίγουρος ότι άκουσα αυτό που μου ζητήσατε, Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι μιλήσατε για τα έργα προτεραιότητας στην Ελλάδα. Ζητήσατε μια ενημέρωση. Μιας και ζητήσατε ενημέρωση λοιπόν για αυτά τα έργα προτεραιότητα στην Ελλάδα, θέλω να σας πω ότι συνολικά είναι πολύ καλή, πολύ θετική η αξιολόγηση για την πρωτοβουλία του Επιτρόπου ΧΑΝ το 2011. Για την Ελλάδα, αυτή η πρωτοβουλία του Επιτρόπου ΧΑΝ έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν έτοιμη να βοηθήσει και αυτή η πρωτοβουλία κινητοποίησε όλους τους φορείς και σήμερα δεν έχουμε μεν την τελική αξιολόγηση. Βλέπουμε όμως ότι τα αποτελέσματα είναι απτά. Από την τελευταία έκθεση που έχουμε για αυτά τα έργα προτεραιότητας, Μάιο του 2017 έγινε η τελευταία αξιολόγηση, και από τα 160 έργα, γιατί κάποια έργα εγκαταλείφθηκαν και βγήκαν από τον κατάλογο, 85% της συνολικής αξίας 7 δισεκατομμυρίων έχουν ολοκληρωθεί, 9% των έργων αυτών, 24 έργα δηλαδή, είναι 770 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν έργα που οργανώθηκαν σε δύο χωριστές φάσεις και θα ολοκληρωθούν στη δεύτερη φάση κατά την τρέχουσα περίοδο και 6% των έργων κόστησαν μισό δισεκατομμύριο. Αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθούν 18 έργα πρέπει να ολοκληρωθούν, διότι είναι μέσα στους, ε, στις διατάξεις μας, πρέπει να ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους μέχρι το 2019. Και αν δεν ολοκληρωθούν μέχρι το 2019, θα ανακτήσουμε την κοινοτική συνεισφορά στα συγκεκριμένα αυτά έργα. Μιας και μίλησα τόση ώρα, Να μην σας πω κι άλλα και σας παρουσιάσω κάποια επιτεύγματα, αλλά είναι τόσο αξιόλογα αυτά τα επιτεύγματα αυτών των έργων που έχουν ολοκληρωθεί και κάποια από αυτά τα επισκεφθήκατε όλες, όπως είπατε. Το δίδαγμα το οποίο αποκομίζουμε από τη διαδικασία αυτή είναι ότι αυτή την προσέγγιση θα την συνεχίσουμε πολύ πιο στοχευμένα και στην τρέχουσα περίοδο με την Ελλάδα. Και προσπαθούμε τώρα με την Ελλάδα να συμφωνήσουμε ένα περιορισμένο κατάλογο, όχι 160 έργα, αλλά πολύ πιο περιορισμένο κατάλογο έργων που θα είναι ιδιαίτερα αξιόλογα και στα οποία θα αποδώσουμε ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Με ρωτήσατε και για το χρονοδιάγραμμα. Τώρα είμαστε στη διαδικασία κλεισίματος. Άρα υπάρχουν προθεσμίες βάσει της νομοθεσίας. Ολοκληρώνουμε τώρα τις παρατηρήσεις μας προς την Ελλάδα, ζητώντας ε, συμπληρωματικές πληροφορίες για διάφορα θέματα. Πληροφορίες και για ορισμένα από αυτά τα έργα από τον κατάλογο προτεραιότητας. Η Ελλάδα θα έχει δύο μήνες στη διάθεσή της μέχρι να απαντήσει στις παρατηρήσεις μας. Θα αξιολογήσουμε τις απαντήσεις και το φθινόπωρο μπορούμε να επανέλθουμε και να σας δώσουμε τα πλήρη και τελικά στοιχεία της αξιολόγησής μας για την έκβαση αυτών των έργων προτεραιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Φθινόπωρο 2017 εννοείται. 2017, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα και θα περιμένουμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις και σίγουρα και οι συνάδελφοι θα έχουν ε, ερωτήσεις. Για τα τέσσερα κράτη-μέλη στο σχέδιο δράσης ε, των ε, κρατικών συμβάσεων, ποια είναι αυτά τα τέσσερα κράτη-μέλη που ακόμη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Μετά Ε, την αποστολή μας είχαμε ασχοληθεί και με τα θέματα αποζημίωσης ε, γεών λοιπά. Δεν ξέρω ε, αν πρέπει όλοι να προσφεύγουν στο δικαστήριο Είμαι μέλος της Επιτροπής ε, παροχής βοηθείας προς την Ελλάδα και αν έχετε κάποια στοιχεία και μπορείτε να μας δώσετε σχετικά με αυτό θα ήταν χρήσιμο. Μπορείτε να μας στείλετε και ως γραπτή απάντηση αν δεν έχετε ε, συγκεκριμένη απάντηση τώρα. Είχαμε ε, κάνει σχετικές συζητήσεις και θα μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι απέγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας που ήταν λεπτομερέστατη. γιατί δεν ήταν τόσο επιτυχής ε, η δράση της προηγούμενης Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιφερειακής Πολιτικής Από αυτά που μας είπατε για τις κρατικές προμήθειες ήταν πολύ, θετικό, θετική αυτή η σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου να δημιουργηθεί ένα μητρό των επιχειρήσεων. Ε, γιατί δεν το ζητά υποχρεωτικά η Επιτροπή από τα κράτη-μέλη και παραμένει ως σύσταση. Είναι ενδιαφέρον να έχουμε την αξιολόγηση ενός έργου ε, σχετικά σύντομα, γιατί τώρα είμαστε στον ΙΣΙΝ 5 νομίζω. Δεν ξέρω γιατί χρειάζεται μια τόσο μακρά διαδικασία για την αξιολόγηση. Και μιλάμε για τα έργα προτεραιότητας, γιατί υπάρχουν και πολλά ε, άλλα έργα στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2014. Η Ελλάδα έχει λάβει αρκετά μεγάλη χρηματοδότηση. Έχετε κάτι να μας πείτε για τα υπόλοιπα έργα που δεν ήταν έργα προτεραιότητας. Αυτές είναι οι δικές μου ερωτήσεις. Και ο συνάδελφος Τσέλα έχει ζητήσει το λόγο. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Η Επιτροπή προσπαθεί να βοηθήσει συγκεκριμένα κράτη-μέλη στην υλοποίηση των ε, προγραμμάτων ε, των έργων του προγράμματος συνοχής. Γίνεται αντίστοιχη συζήτηση και στην περιφερειακή πολιτική. Έγινε και μια συζήτηση με την Επίτροπο Βεστάγκερ για τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων. Υπάρχουν ε, πολλοί ε, κανόνες εξαιρέσεων από ε, τις διατάξεις των κανονισμών. Και η Περιφερειακή Επιτροπή έχει ορίσει τον συνάδελφο Αρεμό ως ειδικό εισηγητή για την Ελλάδα. Την περασμένη εβδομάδα γυρίσει από την Ελλάδα αρκετά απογοητευμένος γιατί είχε επισκεφθεί πολλούς ε, συνομιλητές και δεν είχε σαφή εικόνα για την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Συνοχής. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην χαλαρώσετε την προσοχή σας και να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των έργων της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει και οι χώρες για τις οποίες δημιουργήθηκε το Ταμείο Συνοχής να ξέρουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να επιτύχουν αυτό το οποίο ε, επιθυμούν, δηλαδή δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ε, δημιουργία ανάπτυξης και καλύτερη επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Ευχαριστώ. κυρία Γιάλε Σέντερ. Eh, Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω αν τις τελευταίες μέρες ε, ε, είδατε τα νέα, κύριε ε, Ζέλερ, ότι δηλαδή η Ελλάδα φαίνεται να βγαίνει σιγά σιγά από αυτόν τον κόσμο των ελλημάτων. Ε, ελπίζω σύντομα να ακούσουμε αυτό το καλό νέο και να χαρούμε κι εμείς. Λοιπόν, ε, ήταν καλό το αποτέλεσμα. Τώρα, ε, η Ελλάδα και η υπόθεση της Ελλάδας έχει χρησιμεύσει ώστε να ε, εφευρεθούν ε, μέσα για καλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερα αποτελέσματα. Ε, θέλω να ρωτήσω λοιπόν πρώτον, σε αυτά τα σύμφωνα κυριότητας, ε, ε, ποια είναι η αμοιβή για αυτό τον οργανισμό και κατά δεύτερο λόγο πώς παρακολουθεί η Κομισιόν τα αποτελέσματα. Μετά, για τις απάτες είχαμε δύο διαφορετικές ε, ε, στάσεις. Ε, πώς φτιάχνετε, με ποιες δραστηριότητες μπορείτε να εντοπίσετε τις ύποπτες δραστηριότητες με βάση αυτή τη δράση ε, για τα βασικά αυτά και θεμελιώδη στοιχεία. Αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα. Και τέλος για τις κρατικές ε, ενισχύσεις στο expert group ποιοι ανήκουν και με ποιο τρόπο γίνεται η ad hoc στήριξη. Αν μπορείτε πάλι να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Πυρίνσκι, ευχαριστώ. Έχω κάποιες σύντομες ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Έγινε μια αναφορά στην επίσκεψη που κάναμε το Σεπτέμβριο του 2015. Και από, ως προς αυτό θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι δυνατόν να μας πει η Κομισιόν αν, έχω, αν έχει πληροφορίες για δύο-τρία από τα project, τα έργα που επισκεφθήκαμε. Ένα από αυτά τα project, ένα από αυτά τα έργα που ήταν η δημιουργία κτηματολογίου φαίνεται να έχουν υπάρξει πολλές καθυστερήσεις που οφείλονταν στην έλλειψη ή στην ε, κακή λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού. Οπότε υπήρχε θέμα ε, της αξιοπιστίας των ε, στοιχείων. Και εφόσον αυτό το κτηματολόγιο καθυστερούσε μια ολόκληρη σειρά από άλλα δημόσια έργα και προγράμματα, θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε αν το συγκεκριμένο θέμα το παρακολουθήσατε όλος ιδιαίτερος. Ε, έπειτα υπήρχε ένα πολύ παράξενο έργο ξανα αναζωγόνησης μιας ε, αποξηραμένης λίμνης. Πολύ φιλόδοξο σχέδιο, πρόγραμμα, από μια και από την άλλη η τοπική αυτοδιοίκηση προτίμησε να ε, δημοσιεύσει, την, να δώσει μάλλον δημοσιότητα στη δική μας συνάντηση με τον τύπο παρόντα. Ήθελε λοιπόν να ξαναγεμίσει αυτή τη λίμνη εγκαίρως, γιατί διαφορετικά θα ήταν... Ε, ε, θα καθίσα το γνωστό. Επίσης, άλλο θέμα, το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου κάθε 5-10 μέτρα ένα νέο μουσείο αρχαιοτήτων ε, φτιαχτεί. Ενώ το μετρό δεν έχει ποτέ τεθεί σε λειτουργία ακόμα. Δηλαδή ένα σωρό φιλόδοξα project με αρκετά υψηλό κόστος, τεράστιο αντίκτυπο. Μπορείτε να μας πείτε πού βρίσκονται αυτά όλα. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Είναι το λόγο στον Γενικό Διευθυντή. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρωτήσατε για τα, ποια είναι τα τέσσερα κράτη-μέλη για τα οποία η ολοκλήρωση, η ολοκλήρωση των όρων για τις κρατικές ε, ε, συμβάσεις ακόμα εκκρεμεί. Πρόκειται για τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ιταλία. Η αλήθεια είναι σήμερα ότι η Βουλγαρία είναι σχεδόν έτοιμη. Η Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω. Η Ρουμανία είναι πιο προβληματική. Ε, ε, η κυβέρνηση της Ρουμανίας, η νέα κυβέρνηση της Ρουμανίας αποφάσισε να αλλάξει την προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις και ε, τις στάνταρ δημόσιες συμβάσεις. μόλις πριν λίγες εβδομάδες, πράγμα που μας τοποθετεί σε πολύ αβέβαιη κατάσταση για το πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να συμπεράνουμε, μάλλον καταλήξουμε στο ότι όντως η Ρουμανία έχει ένα πολύ σταθερό και συμβαγές σύστημα δημοσίων συμβάσεων. Έχουμε εντατική επαφή με τις ρουμανικές αρχές και ελπίζουμε ότι αυτό θα καρποφορήσει. Εν καιρό. Ναι. Γιατί όπως είπα, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί να αποφασίσουμε την αναστολή κάποιων ε, πληρωμών μέχρι ότου να τηρηθεί, τηρηθούν οι όροι. Οι ρουμανικές αρχές λοιπόν εργάζονται με εμπειρογνώμονες της ΕΤΕΠ Ο συνάδελφο ε, Νόμανς Πόπεν που τον είδατε και χτες το απόγευμα ήταν εκεί πριν από μία εβδομάδα ώστε να συμφωνήσει ε, στα βήματα που πρέπει να γίνουν ε, στη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί ο χρόνος πιέζει. Εγώ ίδιος θα πάω εκεί το Σεπτέμβριο. Ελπίζω ότι θα μπορέσω τότε να καταλήξουμε, να μπορέσω να καταλήξω στο ολοκλήρωση αυτού, του, αυτής της πρόοδου, ε, πιέζουμε όσο μπορούμε. Αλλά σήμερα δεν μπορώ να πω ότι είναι καθυσυχαστική η κατάσταση για τη Ρουμανία. Είναι πολύ πιο θετική η κατάσταση στα άλλα τρία μέλη στα οποία, τα οποία ανέφερα. Εν γέννη για τους ε, εξάντε όρους φτάνουμε στην ώρα του τελική αξιολογήση, οπότε το φθινόπωρο θα έχουμε αρκετές περιπτώσει να εξετάσουμε γιατί οι εξάντε οροί σχετίζονται και με το περιβαλλοντικό νόμο, για παράδειγμα αν υπάρχει συμμόρφωση με την οδηγία περί υδάτων ή την οδηγία περί αποβλήτων, περί λιμάτων ε, και είναι σαφές ότι ορισμένα κράτη-μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους. Αν όχι, το Σεπτέμβριο θα πρέπει να προβούμε σε κάποια στοχοθετημένη αναστολή πληρωμών. Benefit of this new uh, regulatory frame. Έχουμε δυνατότητα να πιέσουμε τα κράτη-μέλη μέσα σε αυτό το πλαίσιο για τους προσυμφωνημένους όρους ε, εφόσον δεν τους στηρούν. Και πάλι λοιπόν το βλέπω αυτό ως ένα πολύ θετικό μηχανισμό και γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ολοκληρώσουν βελτιώσεις ε, στη, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις λόγω ακριβώς των ε, προσυμφωνημένων όρων και τον ενσωματωμένο μηχανισμό ε, κυρώσεων to, uh, Επίσης ε, θα σας δώσω πληροφορίες γραπτός. γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαι άμεσα ενημερωμένος για αυτό που με ρωτήσατε. Θα σας απαντήσουμε όμως από αυτού. Επίσης, ε, ε, με χαροποιούν οι παρατηρήσεις για τους προκατόχους μου. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι αυτά που σας αναφέρω ε, θα... Μάλλον, ξεκίνησαν υπό τη δική μου αιγίδα. Εγώ ξεκίνησα πολύ αργότερα. Τώρα βλέπουμε τα, τους καρπούς των προσπαθειών των προκατόχων μου. Αλλά θα έλεγα ότι Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα δράσης για τα οποία μιλάμε έχουν φτιαχτεί το 2015, πλέον η πρόοδος είναι ορατή και αρκετά πιστική. Δεδομένου του το, το, το, θέματος μας απασχολεί, είναι το πιο δύσκολο πράγμα νομίζω να το πετύχει κανεί, Δηλαδή η βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων του διοικητικού μηχανισμού. Ε, και κύριε Πυρίνσκι, πολύ σωστά είπατε, αναφερθήκατε σε κάποιες ανησυχητικές εξελίξεις όσον αφορά το κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό δείχνει ε, λήψεις στο λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο να μπορούμε εμείς να διορθώσουμε και σίγουρα δεν διορθώνεται μέσα σε λίγους μήνες. Με το λίγο χρόνο που έχει περάσει από το 2015, σε ε, ενθαρρύνουν τα αποτελέσματα. Έχουμε μπει στο δρόμο, πιστεύουμε. Και ελπίζουμε ότι οι καρποί αυτοί θα πολλαπλασιαστούν σε όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Κεντρικό κτηματολόγιο που ανέφερα, από ό,τι θυμάμαι, το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι της DG ε, ανταγωνισμού. Για τον τελευταίο κανονισμό de η Κομισιόν πρότεινε να είναι υποχρεωτικός ο χαρακτήρας των κεντρικών κτηματολογίων σε εθνικό επίπεδο και τροποποιήθηκε από τον νομοθέτη σε κάτι που ήταν ε, θελοντικό. Αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε κάποια κράτη-μέλη να δεσμευτούν όντως στο να φτιάξουν ε, κτηματολόγιο σύμφωνα με τους ε, προσυμφωνημένους όρους. Δεν μπορούσαμε να τους υποχρεώσουμε γιατί δεν υπήρχε καμία σχετική νομική υποχρέωση. Ορισμένα κράτη-μέλη όμως, ε, συγκεκριμένα η Τσεχία και η ε, Σλοβακία, δέχτηκαν αυτή τη, ανέλαβαν αυτή τη δέσμευση και πλέον έχουν φτιάξει τα εκτιματολογιά τους. On Greek projects για τα ελληνικά ε, ε, έργα, ε, το 160 έργα προτεραιότητας, ναι, θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιονομικών πληροφοριών μόλις θα έχουμε ολοκληρώσει, όπως είπα φέτος, την αξιολόγησή μας. Ρωτήσατε για όλα τα υπόλοιπα στην Ελλάδα, στην ε, πολιτική συνοχής. Εν γέννη, είδαμε πως ε, η Ελλάδα επιτέλους έχει καταφέρει να απορροφήσει όλη τη βοήθεια που ήταν διαθέσιμη μέσω της πολιτικής ε, συνοχής. Αυτό σίγουρα βοήθησε και τώρα αναφέρομαι στο σχόλιο της κυρίας Αγιάλα Σέντερ για να βγει η χώρα και από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Γιατί για όλες αυτές τις αποφάσεις χρειάστηκε να ε, και αυτή η μέθοδος φάνηκε λοιπόν απευχρήσιμη. Δεν γνωρίζουμε κάθε ένα project χωριστά που χρηματοδόθηκε αυτή τη στιγμή ε, μέσω της ε, πολιτικής συνοχής, αλλά πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να σας δώσουμε πλήρη αξιολόγηση για τα τελικά ποσοστά απορρόφησης στην Ελλάδα που θα έπρεπε να ε, είναι γύρω από το 100%. Η Ελλάδα δηλαδή έχει καταναλώσει όλα τα ποσά που τις προσφέρθηκαν. Ε, αλλά ωστόσο συμφωνώ ότι δεν είναι όλα ε, ρόδινα στην Ελλάδα σήμερα. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι στη νέα περίοδο 2014-2020 που η Ελλάδα πρέπει να συγχρηματοδοτήσει ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει το όπως θα θέλαμε. Γι' αυτό και είπα ότι θέλουμε να αποκομίσουμε τα θετικά διδάγματα από την προσέγγιση με την λίστα προτεραιοτήτων, ώστε να μπορέσουμε με πιο στοχοθετημένο τρόπο να συμφωνήσουμε με την Ελλάδα για έναν ε, συγκεκριμένο αριθμό ε, ε, έργων κλειδιών που θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν. Θα, δηλαδή πρόκειται για ένα πιο περιορισμένο κατάλογο 20 με 50 έργων. Πέρα από αυτά όμως θα ε, συνεχίσουμε να συνοδεύουμε την Ελλάδα όσο μπορούμε καλύτερα. Έχουμε κάπως ούριο άνομα, σήμερα γιατί ε, έχουμε αυτά τα project που σας ανέφερα όπου ε, θα χρηματοδοτηθούν ως δεύτερο κύμα έργων με το 2014-2020 αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ότι θα έχουμε την κατάλληλη προετοιμασία για τα επόμενα έργα και εκεί δεν είμαστε ακόμα πλήρως ικανοποιημένοι. Όσον αφορά τα σύμφωνα κεραιότητας που με ρωτήσατε, χρηματοδοτούνται, είναι ιδιωτικά έργα, χρηματοδοτούνται από μέσω της τεχνικής βοήθειας της Επιτροπής. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση εδώ για το μέλλον. Τέτοιου είδους δυνατότητες τεχνικής ε, βοήθειας σε επίπεδο κομισιών είναι απαραίτητη για να δοθεί μια όθηση, εναρκτήρια όθηση σε κάποιες περιπτώσεις είναι για να βελτιωθεί η κατάσταση σε κάποια κράτη-μέλη. Αυτό το, το πολιτικό, πιλωτικό πρόγραμμα Συμφώνου Κεραιότητας χρηματοδοτείται από 11 εκατομμύρια μέσω του προϋπολογισμού τεχνικής βοήθειας που έχουμε σε διάστημα 4 ετών. Θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια και αυτά τα 7 εκατομμύρια ε, είναι στη διάθεση της διεθνούς διαφάνειας οι οποίοι αυτοί θα τρέξουν και θα επιβλέψουν τις διάφορες χωριστές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα εκείνη είναι ο εξωτερικός μας συνεργάτης ο φύλακας, ο θεματοφύλακας της ακαιρεότητας ε, στην στις διαδικασίες αυτή. Και τώρα όσον αφορά τους συμμετέχοντες είναι οι δημόσιες αρχές, ε, οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς, αυτοί που υποβάλλουν προτάσεις, όλοι συμμετέχουν εθελοντικά. Όπως μας δίνει, λέει και το όνομά του, το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα σκοπό έχει να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο την ε, διάδοση, διάχυση αυτού του είδους των ε, έργων στο μέλλον όταν θα μελετάμε την επόμενη προγραμματική περίοδο. Με ρωτήσατε να, σχετικά με τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Ζητήσατε σχετικά συγκεκριμένα παραδείγματα ύποπτων καταστάσεων που θα μπορούσαν να έχουν σχέση με απάτη και που μπορούν να εντοπιστούν μέσω του συστήματος Αράκνη. Καλύτερα να σας στείλω γραπτά την απάντηση. Όμως, το σύστημα είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Σκοπό έχει μέσω της συγκέντρωσης διαφόρων δικτών, δεδομένων να εντοπίζει τις ύποπτες καταστάσεις και συμπεριφορές. Θα λάβετε γραπτή απάντηση. Ο κύριος Μπερίνσκι για το... Ο κύριος Πυρίνσκι για το κτηματολόγιο αυτό νομίζω συζητείται στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Και όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο ε, προς μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας στο μέλλον. Εμείς λοιπόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δω σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το έργο μέσω διαφόρων υπηρεσιών, συνεργασία με την SRSI, την ε, Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Έχουμε στείλει και ειδικούς, από το εξωτερικούς ειδικούς, αν δεν κάνω λάθος, την Παγκόσμια Τράπεζα. Τα χρήματα υπάρχουν, δεν τίθεται θέμα χρημάτων. Τελικά το θέμα είναι οι διοικητικές δομές, η διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Και γι' αυτό σαφώς δεν μπορώ σήμερα να σας πω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πόσο γρήγορα θα εξελιχθούν στο μέλλον. Όμως είναι κάτι που μας ανησυχεί. Και επίσης είναι ένας τομέας που θα, θέ, στον οποίο θα θέλαμε να γίνει ουσιαστική πρόοδος κατά τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής περίοδου. Σίγουρα. Αναφερθήκατε και σε δύο από τα έργα του καταλόγου προτεραιότητας. Τη λίμνη αυτή, η οποία θα αναβιώσει και την οποία είχατε την ευκαιρία να επισκεφτείτε, εγώ όχι. Μου είπαν όμως ότι τα εγγένεια πρόκειται να γίνουν σύντομα. Υποθέτω άρα ότι μέχρι τώρα και πάλι θα πρέπει να έχει εμφανιστεί λίμνη. Ε, τώρα, για, το... για τη Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον επειδή έχει πλούσια ιστορία και προσπαθεί να την ε, διαφυλάξει πολύ σωστά. Το έργο του Μετρό έχει προχωρήσει. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά η κυρία Κρέτσου πήγε και στην, στα εγγένεια ε, ενός τμήματος το οποίο δόθηκε σε λειτουργία. Επ' αυτού λοιπόν δεν ανησυχώ. Ähm, ähm, Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρονται όλα αυτά. Βλέπω ότι δεν ανησυχείτε. Ε, δεν ξέρω αν θα είχαμε προσκληθεί στα εγγένεια. Ε, δεν ξέρω πόσα χρήματα θα χρειαστούν μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση. Χαιρόμαστε για την παρουσίαση και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε άλλη μια σχετική παρουσίαση και μια επίσκεψη στην Ελλάδα. Είδαμε ότι σε όλη αυτή την πορεία Υπάρχει δέσμευση και ενθουσιασμός και δουλειά των ε, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, Ελλάδα. Κανείς δεν αμφιβάλλει από αυτού. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ελλάδα. Μας είπατε το φθινόπωρο. Φθινόπωρο του 17 είπατε. Έχετε και συγκεκριμένο μήνα να μας πείτε ποιο μήνα του φθινοπόρου θα γίνει η επόμενη παρουσίαση θα έχετε ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Σαφώς ε, μας ενδιαφέρει το θέμα της Ελλάδας και με τα χαράς θα σας καλέσουμε για να μας ενημερώσετε κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Σας ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Και την επόμενη φορά θα ήταν πολύ καλό αν είχαμε και αριθμητικά στοιχεία, να έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία που θα μας φέρετε για να μας δείξετε την πρόοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και σας περιμένουμε με την αξιολόγηση το φθινόπωρο. Οπότε, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το υπαριθμό 16 είναι η δική μου γνωμοδότηση για την Eurojust. Θα είμαι σύντομη. Στον κανονισμό της Επιτροπής το θέμα είναι η Eurojust. Υπέβαλε μια πρόταση η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013. Το 2015 εκφράστηκε το Συμβούλιο αφαιρώντας κάποιες διατάξεις που αφορούσαν τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και περίμενε και η Επιτροπή ΛΥΜΕ την έκθεση. Περιμέναμε μέχρι να προχωρήσει και ο κανονισμός ε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα έχουμε την έκθεση και υπάρχει το, θέμα της σχέσης μεταξύ του Ευρωπαίου, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Eurojust. Έχουμε 19 τροπολογίες που χρειάστηκαν αρκετό χρόνο μέχρι να συνταχθούν από τη γραμματεία. Θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό ε, ε, στις σχέσεις ε, με την Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ λέει ότι για όλα αυτά τα οποία δεν είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι αρμοδιότητα της Eurojust. Αλλά έχει και η όλα αρμοδιότητα. Πρέπει λοιπόν τώρα να βρούμε τη σωστή ισορροπία και θα κάτσω και το Σαββατοκύριακο να δουλέψω επ' αυτού για να βρούμε ακριβώς ποια πρέπει να είναι η ισορροπία με τους δύο άλλους οργανισμούς. Η έκθεση ασχολείται με την ε, θεσμική μορφή της Eurojust Προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με τις αρμοδιότητες του διοικητικού διευθυντού προσπάθησα και εγώ και η γραμματεία της Επιτροπής να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Δεν έχουμε καταλήξει στο σύνολο της έκθεσης, αλλά θα κάτσω και το Σαββατοκύριακο, όπως σας είπα, να δουλέψω και ελπίζω ότι τη Δευτέρα θα είναι έτοιμα. 17 Ιουλίου μεσημέρι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Όπως σας είπα θέλει λίγο δουλειά ακόμη. Για αυτό που σας είπα, σχέσεις με Όλαφ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μέχρι τώρα δεν είχαμε προχωρήσει γιατί δεν είχε προχωρήσει και το Συμβούλιο με τον κανονισμό. Και θα κάνουμε και μια συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές όταν έχουμε όλες τις τροπολογίες. Η κυρία Γιάλα Ζέντα έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Διαπιστώνω ότι κάνατε ιδιαίτερη προσπάθεια για να προσεγγίσετε το θέμα Μιλώ εν μέρη τουλάχιστον εκ μέρους κυρίας Χόφμαν, η οποία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. έχουμε κάποια θέματα που μας απασχολούν. Πρώτον, αντί τη δημιουργία ενός EPPO ε, που θα συνεργάζεται με την OLAF αντί να, και τη Eurojust, αντί να μειώσουμε τη γραφειοκρατία ε, αυτό που γίνεται με το νέο σχέδιο κανονισμού αυξάνει η γραφειοκρατία στη Eurojust. Ένα άλλο θέμα που θέσατε κι εσείς είναι η σχέση μεταξύ του νέου EPPO όλα πρέπει να είναι απολύτως σαφέ όταν ε, μιλάμε για τις νέες ε, υποχρεώσεις του, της Όλαφ και της Eurojust. Και μετά τι θα γίνει το ΕΠΠΟ, το, Γραφείο του Ευρωπαϊκού, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα ενισχυθεί και θα λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατόπιν φτάνω στις ε, τροπολογίες. Όσον αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή. Πολύ ωραίο που θα επιβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη θέση αυτή. Θα ήθελα όμως να είναι πιο σαφές. Θα γίνει η ίδια ιστορία όπως όταν πρόκειται για επίτροπο, δηλαδή ακρόαση, κανόνες ε, παρέτησης ή απόλυσης. Ο εκτελεστικός διευθυντής Ε, θα, θα ε, έχει σχέση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι συλλογικό όργανο. Δηλαδή τι θα γίνει, θα είναι μια θέση από διαφομπέου τραγού. Τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν ενδεχομένως θα, θα τον κατηγορούν για τα δικά του σφάλματα. Και όσον αφορά για τον προπολογισμό που δεν είναι και τεράστιος, ναι, ε, ενισχύεται η παρουσία και η ελεγκτική αρμοδιότητα του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά πιστεύω πως, σε πάση περιπτώσει, τις αποφάσεις πρέπει να τις λαμβάνει το συλλογικό όργανο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να απαλλάσσουμε ευθυνών την Κομισιόν που είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. Kollege Κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με δύο λόγια. Θέλω να σας συγχαρώ για την καλή δουλειά που κάνατε και να εκφράσω θερμή υποστήριξη για το γεγονός ότι ασχοληθήκατε ιδιαίτερα με τη διαφάνεια και την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόνων, ως, όπως επίσης και με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Θεωρώ και πάλι ότι αυτά τα τρία θέματα στη, στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης, όπως και σε πολλές άλλες, αποτελούν τα βασικά στοιχεία. Και συνεχίζω, προσβλέπουμε στη συνέχιση της εργασίας. Το θέμα θα το στηρίξουμε στεναρά. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Δεν θέλει κανένας άλλος το λόγο. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε την ε, διοικητική δυνατότητα της Eurojust και όχι να την αποδυναμώσουμε. θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο διοικητικό διευθυντή να εφαρμόζει αυτά τα οποία επιβάλλονται. Όταν υπάρχει μια δομή όπου υπάρχουν πάρα πολλά μικρά τμήματα και δεν υπάρχει μια συνεκτική λειτουργία, αυτό που θέλω είναι να ενισχύσουμε την συνοχή. Υπάρχει όλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Eurojust και η Europol. Υπάρχουν κράτη που είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είκοσι από μια μεριά και 7 από την άλλη. Είναι τέσσερα αυτά τα θεσμικά όργανα που πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδυαστούν. Εφιάλτης πραγματικός. Και συμφωνώ με την ανάλυση της συναδέλφου Αγιάλα Σέντερ. Εγώ προσπάθησα να δώσω ε, ισχυρές εξουσίες. Ε, αν κάνουμε κάτι ε, στο ένα σημείο, επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα σημεία. Αν έχει κανείς κάποια καλύτερη ιδέα, ευχαρίστω, γιατί προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία και ακόμη δεν έχουμε καταλήξει στην ιδανική λύση. Κάθε πρόταση ευπρόσδεκτη. Όπως σας είπα, έχω προβλέψει να δουλέψω το Σαββατοκύριακο πάνω σε αυτό. κυρία Χολμάγερ. Ήταν μακρύς ο δρόμος μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και λυπάμαι που καθυστέρησε τόσο πολύ. Ε, το περιμέναμε σαν κάτι το θετικό και μετά από ε, τόσο μεγάλη πορεία που κάναμε θα τους βγάλει με το δικαστικό κομμάτι. Πρέπει να εναρμονίσουμε τα θέματα της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ της Αγγελίας, Eurojust και Όλαφ. είναι καλό ο συντονισμό τη Eurojust, αλλά παράλληλα υπάρχει και η εισαγγελία που κάνει κάτι άλλο και η Όλοφ που κάνει κάτι ακόμη. Δεν είναι αποτελεσματικό αυτό στο οποίο ε, έχουν καταλήξει τα κράτη-μέλη. Θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό αν χωροταξικά τουλάχιστον τους βάλουμε όλους μαζί στη Χάγη, να μην χρειάζεται να είναι 300 χιλιόμετρα μακριά ένας από τον άλλον. Μέχρι τώρα ό,τι μπορούσε να γίνει λάθος, έχει γίνει λάθος. Από τη Γενική Διεύθυνση Just, η κυρία Μέντρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, της Eurojust και της Όλα. Είναι σημαντικό να είναι σαφής και στο κείμενο η σχέση ε, έχουν γίνει κάποιες τροπολογίες και στην έκθεση της ΛΥΜΠΕ να δούμε αν μπορεί να ξεκαθαριστεί έτσι περαιτέρω η σχέση της Ευρωπαϊκής Αγγλίας με την Eurojust. Όπως είπατε και εσείς, ε, είναι απολύτως απαραίτητο είναι ξεκάθαρο το κείμενο. Τώρα, στο θεσμικό σκέλος, η πρόταση της Κομισιόν συντάχθηκε σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, δηλαδή πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπο της Κομισιόν στο Διοικητικό και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Δεν έχετε κάνει αλλαγές εκεί, αλλά η έκθεση ΛΥΜΠΕ επέκλεισε την Κομισιόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί η Κομισιόν και χαίρομαι που εσείς ε, συμφωνείτε μαζί σας, γιατί όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό να είναι σε αυτό το Συμβούλιο η ε, Επιτροπή Τώρα, όσον αφορά την ε, ε, επιλογή του διοικητικού διευθυντή, ε, η Επιτροπή θα κάνει την επιλογή των υποψηφίων και ο σύντομος κατάλογος θα υποβληθεί στο Συμβούλιο. Δεν συναναφέρεται αυτό στην έκθεση της ΛΥΜΠΕ, όπου δεν αναφέρεται αυτό. Αλλά πιστεύουμε ότι και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει και βλέπουμε ότι και εσείς και σε αυτό μας έχετε υποστηρίξει. Αυτή είναι η μόνη παρατήρηση, το μόνο μου σχόλιο.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 Όπως είπαμε, αν υπάρξουν σχετικές προτάσεις, ε, ε, τις αναμένουμε. Υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούσε να ακουστεί η διερμηνία. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τα σημεία της σημερινής διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το σημείο αυτό, επαναλαμβάνω, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. 4 Σεπτεμβρίου θα ασχοληθούμε και πάλι με το θέμα αυτό και θα προσπαθήσω να οργανώσω μετά τις καλοκαιρινές διακοπές ε, μια συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τους σκιώδεις εισηγητές ε, να το συνδιαμορφώσουμε. Λοιπόν, όπω είπαμε, ολοκληρώσαμε την σημερινή μα συνάντηση. Θα ακολουθήσει μια σύντομη συνάντηση των συντονιστών. Καλέ διακοπέ ε, και να γυρίσετε κεφάτη και υγιείς. Όσοι δεν συμμετέχουν στη συνάντηση των συντονιστών, παρακαλώ σύντομα να αποχωρήσουν.